Allora, riprendiamo i lavori. Ehm, cominciamo dal terzo cluster. Dal titolo... Να περάσουμε στο τρίτο κλάστερ, να διερευνήσουμε τους τρόπους για να βελτιώσουμε τις ενέργειες και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμών, των υπηρεσιών και τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται ε, στην, ε, στον εντοπισμό και στην καταστολή της ε, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Λοιπόν, θα έχουμε 15 λεπτά χρόνο για τον καθομιλητή και κατόπιν θα κάνουμε τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τη Σοφία Συνπέρο από την ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών για τη συνεργασία των τραπεζών με ε, τις μονάδες διοικητικών υπηρεσιών και τις διοικητικές αρχές. Κατόπιν θα μας μιλήσει ο για το ρόλο... Ε, του Ιδρύματός του για την συνεργασία και θα μας μιλήσει για τις ε, συνέργειες και την συνεργασία ε, στις διοκτικές αρχές που σχετίζονται με το ξέπλυμα βρώμικου Θα ξεκινήσουμε με τη Σοφία Συντερό για 15 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτέ. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να παρουσιαστώ ενώπιον σας σήμερα. Ο κύριος Αρή Καντάρ προβλεπόταν να μιλήσει σήμερα, αλλά δυστυχώς είχε ενηλυμένη υποχρέωση της τελευταίες στιγμής. Γι' αυτό θα είμαι σύντομη. Θα σας παρουσιάσω την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία που θέλει να είναι η φωνή των ευρωπαϊκών τραπεζών εκπροσωπούμαστε σε 31 χώρες, τις 27 της Ένωσης, τις 4 της ΕΖΕΣ και 4.000 τράπεζες με 5.000 υπαλλήλους. Εκπροσωπώ λοιπόν μία ομοσπονδία που η ίδια εκπροσωπεί τις τράπεζες. και έχουμε και εμείς μια άποψη για τη συνεργασία των τραπεζών με τις κυψέλες ή κύτταρα δημοσιονομικής πληροφόρησης. Ιδίως για την καταπολέμηση των φαινομένων ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος. Και σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα αλλά και το γενικότερο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Στο ένα πρώτο μέρος της παρουσίασής μου θα υπενθυμίσω ποιες ήταν οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει για την καταπολέμηση μεταξύ άλλων της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα πιστοτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών και πελατριών τους, σωματική και ηθική, για να είναι βέβαιοι για την ε, εμπορική τους ε, δραστηριότητα. Αυτά όλα τα γράφουμε ηλεκτρονικά ή σε χαρτί και τα πιστοτικά ιδρύματα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά τις πληροφορίες αυτές. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε τον πελάτη, δηλαδή τα πρόσωπα που έχουν πάνω από 25% μετοχών σε μία τέτοια ηθική ταυτότητα. Οι πελάτες υψηλού κινδύνου όπως οι όσοι εκτίθενται σε πολιτικούς κινδύνους όπως εσείς κυρίες και κύριοι βουλευτέ, όσοι δηλαδή όσα φυσικά πρόσωπα έχουν δημόσια δραστηριότητα. Γι' αυτό λοιπόν ε, υπάρχουν εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου ή μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου που γίνονται και ανθρωπίνος με κάποιον αξιωματούχο και υλικός, δηλαδή με τη χρήση τεχνολογίας. Τα περισσότερα ιδρύματα χρησιμοποιούν αυτόματα συστήματα καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι ύποπτες δοσοληψίες πρέπει να δηλώνονται αρμοδίως και να γίνεται ανάλυση και αν χρειάζεται να αναφέρεται στις αρχές το συμπέρασμα. Αν υπάρξει συμπέρασμα δηλαδή για ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος. Υποχρέωση λοιπόν πληροφόρησης και ενημέρωσης. Τα ιδρύματα αυτά έχουν μεγάλη πείρα και στην καταπολέμηση τέτοιων δοσοληψιών και στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τις μονάδες ε, χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης έχουμε ένα έντυπο που σας το επέδειξα εδώ από το 2008 που δείχνει ότι 80% των σχετικών δηλώσεων προέρχονται από χρηματοπιστωτικά ιδουρήματα. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και με τις τράπεζες στο πλαίσιο της υποχρέωσης πληροφόρησης που έχουν οι μονάδες που σας είπα. Επίσης μπορούμε να παγώσουμε λογαριασμούς και να επιτηρήσουμε διαμεθοριακές δοσοληψίες όπως συστήνει η σύσταση 16. Αυτό ήταν το γενικότερο πλαίσιο των υποχρεώσεων των τραπεζικών ή τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών τυγούτων και τώρα θα σας πω πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν όλα αυτά ακόμη περισσότερο. Πρώτον, καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες δημόσιου χαρακτήρα. Σας είχα πει ότι υπάρχει υποχρέωση να γνωρίζουμε τον πελάτη μας αλλά η τράπεζα τελικά εξαρτάται από αυτά που δηλώνει ο πελάτης. Για να γνωρίζουμε λοιπόν καλύτερα τον πελάτη και την πελάτησα, πρέπει να γνωρίζουμε και ποιοι ακριβώς είναι οι μέτοχοι των επιχειρήσεων. Άρση φραγμών, νομικών φραγμών που μπορεί ακόμη να υπάρχουν για την ε, χορήγηση πληροφοριών μεταξύ περιφερειών ή χωρών θα ήταν επίσης μια βελτίωση. Αυτό το λέω γιατί ξέρω ότι οι ορισμένα μέλη της Επιτροπής σας αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται την αναθεώρηση του γενικότερου πλαισίου προστασίας των δεδομένων και γι' αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων καταπολέμησης της ξεπλήματος δρομικού χρήματος. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει θέμα με την υποχρέωση πληροφόρησης un banquier gère par nécessité des για ορισμένα πρόσωπα για την καταπολέμηση πιθανών απατών, ε, χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Υπάρχουν ορισμένες νομικές ρήτρε για την προνομιακή πληροφόρηση ορισμένων και μοιημένων. Πρέπει οι τράπεζες λοιπόν να ταυτίζουν τον πελάτη ή την πελάτησα, αλλά και κάθε πρόσωπο που έχει ορισμένες τυχές ή όχι σταθερές δοσοληψίες αν ξεπερνάει το ποσό τα 15.000 ευρώ. Είναι υποχρεωμένη η τράπεζα για πέντε χρόνια να διαθέτει τις πληροφορίες για αυτά τα πρόσωπα. Και πρέπει να καθορίζουν επίσης αν ο πελάτης έχει πολιτική έκθεση. Είναι λοιπόν θεμητό ότι οι τράπεζες οργανώνουν ε, τράπεζες δεδομένων για τα πρόσωπα αυτά για να γνωρίζουν και με ποια πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα ή δεν θέλουν να έχουν δοσοληψίες. Πρόσωπα που έχουν μη λευκό ποινικό μητρό ή έχουν δηλωθεί non grata από την Ένωση η καταπολέμηση του πλησίματος μαζί με την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο να διασφαλιστεί. Στον νέο ορισμό της λέξης συνένεση για την προστασία των δεδομένων η συνένεση δεν μπορεί να είναι σιωπηρή, πρέπει να είναι ρητή. και να εκφράζει τη συμφωνία του ενδιαφερόμενου για την χορήγηση των προσωπικών του δεδομένων και την επεξεργασία τους. Μόνο με αυτή τη συνένεση γίνεται. Υπάρχει η δυνατότητα να γνωστοποιηθεί το όνομα κάποιου, αν ζητήσουμε την άδειά του δηλαδή. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει ότι σε περίπτωση που υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε, ένα, σε μια τράπεζα δεδομένων όπως σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο δεν χρειάζεται η συνένεση. Πάντως, αν υπάρχει το όνομα κάποιου σε μια δική μας τράπεζα δεδομένων σημαίνει ότι έχει ήδη δεχτεί. Και ότι όλα αυτά έχουν συλλεχθεί με τον δέοντα τρόπο. Με βάση το νέο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων απαιτείται απλοποίηση και δεν θα υπάρχει πια στο εξή η λέξη διαβούλευση των δεδομένων ή συμβούλευση. Να δεν μπορεί κανείς να συμβουλευτεί τα δεδομένα αυτά. Άλλο θέμα στη συνεργασία με τις μονάδες πληροφόρησης είναι η ομοιομορφία που απαιτείται. Δηλαδή μια τράπεζα πρέπει να δηλώνει, για να δηλώσει ότι μια δοσοληψία είναι ύποπτη, πρέπει να συμπληρώνει το σχετικό έντυπο. Και διαπιστώσαμε στο Λίξεμβούργο ότι μπορεί και ηλεκτρονικά να συμπληρώνεται το σχετικό δελτίο ή έντυπο και στα αγγλικά. Υπάρχει βέβαια το θέμα του εμπιστευτικού χαρακτήρα, του απόρριτου δηλαδή για τις πληροφορίες αυτές. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, ένα πραγματικό feedback και παρακολούθηση των αστυνομικών ερευνών χρειάζεται. Η καταπολέμηση του πλησίματος κεφαλαίων και της τρομοκρατίας μπορεί να γίνει και με συνδυασμό των υπαρχόντων στατιστικών στοιχείων και γι' αυτό υπάρχει ένα εργαλείο και ένα feedback γενικότερο, αριθμούς και δεδομένα, ονόματα για τις ύποπτες δασαληψίες. Η συνέχεια που δίνεται σε τέτοιου είδους δηλώσεις, σε αιτήσια βάση, πόσες υποθέσεις έχουν σημειωθεί, πόσοι καταδικάστηκαν, πόσοι κατηγορήθηκαν, πόσοι λογαριασμοί πάγωσαν, πόσες κατασχέσεις έγιναν και πιο συγκεκριμένα πρόσωπα. Ορισμένες χώρες μέλη τα κάνουν όλα αυτά, αλλά γενικά ατύπως για να μην ε, τεθεί εν κινδύνο κάποια έρευνα ή για να προστατευτούν τα προστατευτικά δεδομένα ή γιατί δεν υπάρχουν επαρκή πόροι για να γίνει η έρευνα. Η αναθεώρηση της τέταρτης οδηγίας κατά του πλησίματος στο... πρέπει ακόμη να καθορίσει σαφέστερα τι εννοεί ακριβώς η έννοια του feedback. Αριθμός ερευνών πόσες φορές έχει επιτυχώς γίνει μια έρευνα κτλ. Η μελέτη λοιπόν αυτή της Κομισιόν από το 2008 για το feedback αυτό συνοψίζει νομίζω πολύ καλά τα πράγματα και διαβάστε τα όλοι. Εξάλλου οι τράπεζες πρέπει να επιμορφώνουν και το προσωπικό τους για να αναγνωρίζουν τα ίχνη και τις ενδείξεις πλησίματος και γι' αυτό χρειάζεται τακτική ενημέρωση των μεθόδων και έμεση δείκτες βέβαια και ενδείξεις. Άρα η πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα των σχετικών ερευνών είναι κάτι το ουσιώδες αν δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ερευνών, του reporting μας δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αποτέλεσμα. Θα γίνονται όλα σαν ρουτίνα που χωρίς ένα νόημα. Ενώ εμείς θέλουμε οι υπάλληλοι των τραπεζών να έχουν συνείδηση των πιθανών κινδύνων και να τους γνωρίζουν. Για να δω αν μπορώ να συμπεράνω τώρα τίποτα η συνεργα... στενή συνεργασία ενισχυμένη μεταξύ τραπεζών και μονάδων δημοσιονομικής πληροφόρησης καθώς και διοικητικών αρχών είναι κάτι το ουσιώδες για να καταπολεμηθεί το πλήσιμο βρωμίκου χρήματος και η χρηματοδότηση της τραμακρατίας. Χρειάζεται συνεννόηση και να συμπερίσσονται όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν γιατί όλοι μαζί έχουμε το κλειδί για να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και να εμποδίσουμε το πλήσιμο και την τρομοκρατία. Δεν μπορούμε βέβαια να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία και με τους άλλους. Τελεία. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ραφέλ. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως αυτή την δική επιτροπή που με κάλεσε εδώ. Συνήθως ε, δεν συνηθίζεται να καλείτε ε, κάποιον ε, που ασχολείται πρακτικά με τα ζητήματα και μάλλον κάποιος σαν και εμένα, αλλά εγώ έχω εμπλακεί σε όλες τις πτυχές τέτοιων εγκλημάτων διαφθοράς από δημοσίους υπαλλήλου για 25 χρόνια και κυρίως ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από τότε που εισήχθη η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1986 και κατόπιν με θέματα όπως ε, η φοροδιαφυγή και η διαφθορά. Και φυσικά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία συζητείτε, συζητάτε εσείς. Θα με συγχωρήσετε αν προσεγγίσω το θέμα με ένα γενικό τρόπο γιατί νομίζω ότι αν έχω κάποια συνεισφορά να κάνω στις συζητήσεις σας είναι στη βάση του να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας και την πρόσφατη αλλά και την πιο μακρινή και να παράσχω συμβουλές όπως έχω κάνει και στο παρελθόν. Έχω δώσει συμβουλές σε άτομα, σε κυβερνήσεις ε, και σε οργανισμούς τα τελευταία 25 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που έχουμε τέτοιους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανομών Όπως ξέρετε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως και αλλού ο κανονισμός για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο ε, και η επιβολή κυρώσεων ε, είναι κάτι προοδευτικό, ένα προοδευτικό εγχείρημα που ξεκινά με την καταπολέμηση της έλευσης ε, του οργανωμένου εγκλήματος ε, που ασχολήθηκε με διακίνηση ναρκωτικών και κατόπιν ασχολήθηκε και επεκτάθηκε σε, ε, με τρομοκρατικές πράξεις, όπλα μαζικής καταστροφής και στη συνέχεια με, με φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα και το οργανωμένο αλλά και το μη οργανωμένο και θέλω να σταματήσω μια στιγμή εδώ και να σας πω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στο επικεντρωνόμαστε μόνο στο οργανωμένο έγκλημα, όπως και αν το ορίζεται και όπως και αν ορίζεται από το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει ένας κίνδυνος ότι άλλα είδη αρκετά σοβαρού οικονομικού εγκλήματος δεν θα αντιμετωπιστούν πλήρως, γιατί το οικονομικό, συγγνώμη, το οργανωμένο έγκλημα προϋποθέτει ότι πρόκειται να υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία μεταξύ ενός αριθμού ατόμων ε, είτε σε μία συστημένη συμμορία είτε σε ένα δίκτυο ad hoc. Αλλά φυσικά αν ε, ασχοληθείτε με θέματα όπως η διαφθορά δεν ε, υπάρχουν πάντα τα συμπτώματα του οργανωμένου κλίματος σε τέτοια περίπτωση και αν μιλάμε για αρκετά σοβαρές απάτες πολύ συχνά δεν λαμβάνουν υποθέσεις αυτές τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι πιο πιθανό να δείτε ε, τα ε, έσοδα που προέρχονται από τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό το έγκλημα να ξεπληθούν ε, σε κάποιες τράπεζες, παραδείγματο χάρη. Το πρόβλημα με τον έλεγχο του εγκλήματος σε όλο αυτό το τομέα αναδεικνύεται καλύτερα από την ε, εισαγωγή νόμων για την καταπολέμηση ε, του ξεπλήματος όταν εισήχθησαν. Γιατί όταν εισήχθησε αυτή η νομοθεσία σήμαινε ότι η υπήρξε αναγνώριση ότι είχαν αποτύχει οι συμβατικές μέθοδοι καταπολέμησης του φαινομένου, γιατί το έγκλημα είχε γίνει διασυνοριακό, είχε περάσει τα σύνορα και ξεπερνούσε τις πολιτικές και τους νόμους των κυρίαρχων κρατών και φοβάμαι ότι αυτό το ε, αίσθημα της απελπισίας που ένιωθαν οι κυβερνήσεις όταν ε, συζητούσαν αυτό το θέμα το 1980, τη δεκαετία του 80, αυτό το αίσθημα της απελπισίας ε, συνεχίζει να υπάρχει σήμερα. Θεωρώ ότι όλο ένα και περισσότερες πολιτικές δημορφώνονται όχι μόνο εδώ, στο επίπεδο Ευρώπης, αλλά και στα κράτη εκπονούνται πολιτικές ε, που προσπαθούν ε, να καλύψουν όλο το σύστημα της συνεργατικής δικαιοσύνης. Δηλαδή και η κοινωνία προσλαμβάνεται σε διάφορες μορφές της για να βοηθήσει τις διοκτικές αρχές. Και πολλές φορές φαίνεται σαν να αντικαθιστά και τις διοκτικές αρχές. Και θα πρέπει να το έχει αυτό κάποιο κατά νου. Μπορεί να είναι αναπόφευκτο, αλλά νομίζω όταν ε, δημιουργείται κάποια μέσα για να την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων όταν καταρτίζετε τα νομοθετήματα πρέπει να έχετε κατά νου ότι τα παραδοσιακά μοντέλα αστυνόμευσης με τα οποία πολλοί από εμά μεγαλώσαμε μερικές φορές ε, είναι εντελώς άσχετα γιατί η συνεργατική δικαιοσύνη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ε, καταγγελία από τρίτο μέρη, αλλά και στην αυτοκαταγγελία, στην αυτοαναφορά. Αυτά που λέω εγώ πρέπει να ειδωθούν υπό αυτό το πρίσμα. Γιατί αν περάσετε νόμους που προϋποθέτουν το παλιωμοδίτικο μοντέλο, ότι θα υπάρχει δηλαδή ένας νόμος που θα επιβληθεί μέσω της έρευνας και θα υπάρξουν πραγματικά αποτρεπτικές κυρώσεις, αυτό το μοντέλο φοβάμαι είναι παροχημένο γιατί οι χώρες δεν έχουν τους πόρους ε, να κάνουν συμβατικές έρευνες. Πρέπει να βασιστούν στο ότι θα τους παράσχονται πληροφορίες και μερικές φορές ότι θα τους δοθεί και όλη η υπόθεση. Η έρευνα, οι μαρτυρίες, οι στόχοι. Ακόμη και ανείχνευση περιουσιακών στοιχείων συνήθω γίνεται από την κοινωνία των πολιτών πριν να μπορέσουν να φτάσουν και οι διοκτικέ αρχέ. Και σε πολλέ περιπτώσει σήμερα οι διοκτικέ αρχέ δεν απασχολούνται καθόλου ή αν ε, έρθουν σε επαφή με τι ιδιοκτικέ αρχέ, δεν έχει τα μέσα η διοκτική αρχή να αντιμετωπίσει το θέμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η δική μας ε, πόροι περιορίζονται, μειώνονται για οικονομικούς λόγους. Η αστυνομία χάνει το 20% των πόρων της. Και οι κυβερνήσεις αναμένουν από τις υπηρεσίες τους διοκτικές να κάνουν περισσότερα με λιγότερο. Επομένως, αν πρόκειται να αντικαταστήσετε ένα μοντέλο, με ένα άλλο, τότε θα πρέπει να πάρετε μαζί σας τους συνεργάτες, θα πρέπει να πάρετε μαζί σας την κοινωνία των πολιτών και προκειμένου να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να δείτε πώς εφαρμόζονται οι νόμοι σας με έναν τρόπο που να πείσετε την κοινωνία των πολιτών. Γιατί σε αυτό θα πρέπει να βασιστείτε περισσότερο στο μέλλον. Θα πρέπει να πείσετε την κοινωνία ότι τα μέτρα που εισαγάγονται είναι λογικά αναλογικά και δίκαια. δίκαια. Όχι μόνο στη σύλληψή τους, αλλά και στη διαδικασία. Και για τη διαδικασία θέλω να πω δύο λόγια. Η προηγούμενη ομιλήτρια μίλησε για τις τράπεζες. Εγώ δεν έχω πολλά να πω για τις τράπεζες, εκτός από το ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο αν ε, και υπήρχαν πρόσφατα κάποια σκάνδαλα πολύ γνωστά με τις τράπεζες, ε, δεν υπήρξαν διώξεις μεγαλών τραπεζών. Αν ε, έγινε αυτή η διαδικασία του name and shame, δηλαδή τις ονόμασαν και τις ντρόπισαν, αυτό έγινε μόνο δικαιτικά, αλλά όχι ποινικά. Αλλά... Υπήρξαν κάποιες έρευνες, αλλά τελικά Όσοι ασχολούνται με την επιβολή του νόμου, όπως εγώ, προβλέπουν ότι θα υπάρξουν διώξεις, αλλά μάλλον κατά ατόμων και όχι κατά θεσμών. Και φυσικά είναι πολύ απλή απάντηση. Καμία αναπτυγμένη κοινωνία ή οικονομία δεν μπορεί να καταστρέψει το τραπεζικό της σύστημα. Αν αφαιρέσουμε μία άδεια από μία μεγάλη τράπεζα, δεν είναι μία πραγματική επιλογή. Διαφορετικά θα φτάσουμε στην ίδια κατάσταση όπως έγινε με τον Άνθρανα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αδίκως ε, κατηγορήθηκε και παρόλα αυτά καταστράφηκε όλη η λογιστική πρακτική τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας επισημάνω είναι ότι οι τράπεζες που παρέχουν λιανικές υπηρεσίες δεν ασχολούνται καθόλου με τη μεταφορά μικρών ποσών μικρών χρηματικών ποσών. Δεν ασχολείται με αυτό γιατί ο κίνδυνος, δηλαδή η ανταμοιβή, δεν ε, είναι λογική. Είναι πάρα πολύ ψηλή η κίνδυνη και μάλλον ε, δεν υπάρχει κάποιο ε, κέρδος για τις τράπεζες. Όμως το Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες εργαζομένους οι οποίοι αναπόφευκτα στέλνουν ένα τμήμα ή όλο το μισθό τους πίσω στην πατρίδα τους. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο όγκο ε, κυκλοφορίας μικροποσών που σε κάποιο στάδιο πρέπει να μπουν σε κάποιο διεύλο και ο διεύλος που χρησιμοποιείται είναι ε, κάποιοι οργανισμοί, κάποιες επιχειρήσεις που στέλνουν χρήματα και αυτό γίνεται ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Έχει αναγνωριστεί ότι αυτά τα γραφεία είναι πρόβλημα. Τα έχουμε ρυθμίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2003 αλλά είναι διαφόρων μεγεθών. Έχουμε τεράστια τέτοια γραφεία όπως η Western Union και έχουμε κάποια μικρότερα ε, όπου απασχολούνται ένα-δύο άτομα και εκεί προσφεύγουν κυρίως μετανάστες ή εθνοτικές ομάδες για τις υπηρεσίες τους και φοβόμαστε ότι θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κανάλια από το οργανωμένο έγκλημα για να διοχετεύσουν ε, τα προϊόντα του εγκλήματο. και είναι αιτιολογημένο αυτός ο φόβος, Απλώ δεν το ξέρουμε. Αν μπορώ να αναφερθώ σε ένα σχόλιο που έγινε από την προηγούμενη ομιλήτρια που έχει να κάνει με το feedback. Όλοι πάντοτε συζητούν τα μέτρα κατά πολέμηση νομιμοποίηση παρανομισόδων και τελικά καταλήγει σε αυτό το θέμα του feedback. Γιατί? γιατί η τραπεζική κοινότητα και οι υπηρεσίες αυτών των γραφείων και οι διαβαστές πληρωμών ε, ουσιαστικά ε, ζητάνε να τους πούν ε, να τους δώσουν πληροφορίες. Ο, υπάρχει όμως έλλειψη βούληψης από τις διεκτικές αρχές να δώσουν πληροφορίες γιατί μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο οι έρευνες. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία λοιπόν εδώ. Τώρα, η... εγώ δεν θέλω να... δεν εκπροσωπώ εδώ σε καμία περίπτωση ε, τις υπηρεσίες δεκίνησης χρήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, εδώ κάνω κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις, ούτε κάνω να τις ε, σχετίσετε με το δικηγορικό μου γραφείο. Επομένως, όταν ε, σας λέω, ναι, σκεφτείτε το πώ να βελτιώσετε τα πράγματα, αλλά αν κάτι πρέπει να κάνετε είναι να καταστρέψετε τον κινησμό στην κοινωνία των πολιτών που πιστεύει ότι οι περισσότερες από τι ρυθμίσει, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουμε περίπου ε, νομίζω 280.000 ε, αναφορές για ύποπτες συναλλαγές και αν ε, τύχουν επεξεργασίας ε, θα υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει το αφαιρέτο feedback για να δούμε πόσο παραγωγική ήταν όλη αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει μια κοινική άποψη τώρα ότι με την οικονομική κρίση πολλές από αυτές τις πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν απλώς ε, για να διωχθούν οι φοροδιαφεύγοντες και για την ανάκτηση των φορολογικών εσόδων, παρά για το αρχικό στόχο για να καταπολεμήσουμε αυτό το μεγάλο κακό το σοβαρό έγκλημα. Όταν ε, ε, μιλάμε ε, για έρευνα που, που καταλήγει σε κάποιες βλάβες, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όμως, όλες αυτές οι πληροφορίες, ε, νιώθει οι άνθρωποι ότι αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Πρέπει όμως ε, ε, οι ιδιοκτικέ αρχέ να πείσουν του πολίτε ότι αυτή δεν είναι η κύρια χρήση. Είναι μια νόμιμη χρήση, αλλά δεν είναι η κύρια χρήση. Αυτά ήθελα να πω. Όσοι με έχετε ξανακούσει να μιλάω, αυτό είναι ο πιο σύντομο λόγο, η πιο σύντομη ομιλία που έχω δώσει και θέλω να σα καθησυχάσω. Ευχαρίστω να απαντήσω σε ενδεχόμενε ερωτήσει ε, στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε που σεβαστήκατε το χρόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρίγκο, 15 λεπτά και για σας και κατόπιν θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Right. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας απευθύνω το λόγο. Είναι πάντα χαρά το να μπορεί κανείς να μιλάει στο ίδιο βήμα με τον ε, κύριο Ραφαέλ ε, και πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά που είπε και σε ορισμένα θέματα, σε ορισμένα σημεία θα διαπιστώσω ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων. Θα το δείτε εντός ολίγου. Νομίζω γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο εκτελεστικός γραμματέας της Μανιβάλ ε, που είναι ο ε, ελεγκτικός βραχίωνας του Συμβουλίου της ε, Ευρώπης ε, στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Συμμετέχω σε αυτό το μηχανισμό ε, με βάση τη σύμβαση του 2005 για την οποία θα σε ενημερώσω εντό ολίγου γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σύμβαση ε, στο πλαίσιο του νομικού οικοδομήματος της Ευρώπης. Όσον αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης, κοιτάξτε, το Συμβούλιο της Ευρώπης δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Μάλιστα, το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν ο πρώτος οργανισμός που ε, ασχολήθηκε με τους κινδύνους που ελοχεύουν ε, στο βρώμικο χρήμα, σχετικά με το βρώμικο χρήμα και ο λόγος είναι ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με νομικές δεσμεύσεις και είναι ο πρώτος που επιλήφθηκε του ξεπλήματος όπως σας είπα και αυτό διότι το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι για να έχουμε αποτελεσματικό αγώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί από αποτελεσματικά το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Το οργανωμένο έγκλημα είναι, δραστηριοποιείται ιδιαίτερα, πολύ ενεργό, πολύ κερδοφόρο στην Ευρώπη. Και επίσης ε, θέλω να επισημάνω αυτά που είπε ο κύριος Ραφαέλ ε, σχετικά με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ε, μερικές φορές, ορισμένες περιπτώσεις, να τις ταυτίσει κανείς με οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν εγκληματίες ε, οι οποίοι ε, κερδίζουν τα προστοζήν αποκλειστικά και μόνο από το έγκλημα. Και η κοινωνία των πολιτών πρέπει λοιπόν να έχει κάποια σιγουριά ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα εντοπιστούν και αυτοί αλλά και οι άλλοι που τους δίνουν τη δυνατότητα να ε, διαφυλάξουν τα κέρδη τους και αυτοί θα διωχθούν. Σήμερα το 2012 θέλω να πω ότι το να αντιμετωπίσει κανείς ε, το κερδοφόρο έγκλημα, το έγκλημα που αποφέρει κέρδη, αυτό από πλευράς ε, εφαρμογής και επιβολής του νόμου σημαίνει παρακολουθεί κανείς ε, τα κέρδη σε πολλές περιπτώσεις και αυτό παράλληλα με, την, με τις κανονικές έρευνες της αστυνομίας που διεξάγονται για, την, για τον εντοπισμό των αυτούργων. Αυτές οι οικονομικές ε, ανακρίσεις είναι εκείνες που οδηγούν στον ε, εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων ξεπλήματος. Ε, σας λέω, μιλάμε για σοβαρές περιπτώσεις που θεωρώ ότι είναι η ουσία του προβλήματος με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να φτάσει και στα κέρδη τα οποία είναι δυνατόν να κατασχεθούν. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα ε, σωστό ε, νομικό σύστημα, ε, διατάξεις που να εφαρμόζονται και κυρίως νόμοι οι οποίοι θα επιτρέπουν να εντοπίσει κανείς, να κατάσχει και να δημεύσει τα κέρδη. Δεν εννοώ απαραίτητα τα άμεσα, αλλά περισσότερο τα έμεσα κέρδη. Δηλαδή τα σκάφη, τις βίλες, τα χρήματα που έχουν επενδυθεί. Αυτά λοιπόν είναι ορισμένα από τα θέματα που αποτελούν την ομπρέλα του, ε, της συζήτησης μας σήμερα. Εξετάστηκαν και από τον κύριο Ραφαέλ αυτά σήμερα. Έτσι λοιπόν το 2012 για να γίνουν όλα αυτά ε, χρειάζεται να, υπάρχει, να υπάρχουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις νομικής αρρωγής, κυρίως για τον εντοπισμό, το πάγωμα και την ε, κατάσχεση των ε, κεφαλαίων που κινούνται ανά τον κόσμο. Η Μάνεβαλ έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο και συμμετέχει, όπως σας είπα, στο πλαίσιο της Σύμβασης του 2005. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται το δικό της το νομικό οικοδόμημα για να στηρίξει όλα αυτά τα θέματα με αποφάσεις πλαίσιο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σχετική οδηγία σχετικά με τις κατασχέσεις. Πολύ καλά όλα αυτά και λειτουργούν αποτελεσματικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το μήνυμα που θέλω εγώ να εκπέμψω σήμερα το απόγευμα και είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη είναι ότι το έγκλημα, κυρίως ε, το διεθνές ε, έγκλημα, δεν αρχίζει αλλά ούτε και τελειώνει στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει δηλαδή, πολύ σκληρά για να αυξήσει ε, τις εξουσίες για τη διεξαγωγή ερευνών που έχει, αλλά παρεμφερείς εξουσίες πρέπει να δοθούν και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να απευθύνονται σε κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη στο Βέλγιο, παραδείγματος χάνει το Βέλγιο και η Λετωνία, να μπορούν να απευθυνθούν στην Ουκρανία που έχει ε, προσυπογράψει μία από τις συμβάσεις μας. Με τον ίδιο τρόπο που ε, θα μπορούσε κανείς να απευθυνθεί και σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικά θέματα στον αγώνα ε, κατά του υπερεθνικού ε, εγκλήματος, οργανωμένου εγκλήματος. Θα επανέλθω σε αυτό εντός ολίγου. Τώρα, θα ήθελα να πω και λίγα λόγια σχετικά με την ε, Moneyval. Η Moneyval ιδρύθηκε το 1997 την επόμενη εβδομάδα θα ερτάσει την 15η επέτειό της. Αρχικά συσταθήκαμε για να καλύπτουμε εκείνα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, που δεν είναι μέλη της ε, Task Force. Ε, μερικά από τα μέλη μας ήρθαν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και συζήτησαν μαζί σας. Δηλαδή συστηθήκαμε για να καλύψουμε αυτό που τότε το 1997 ε, αποκαλούσαμε τα κράτη σε μετάβαση. Ε, τώρα ε, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλη μια η Κροατία πρόκειται να ενταχθεί την επόμενη χρονιά. Είμαστε τώρα υπεύθυνοι για 33 ε, νομολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα το Συμβούλιο των Υπουργών δέχθηκε την αίτηση του ε, Ηνωμένου Βασιλείου να είμαστε αρμόδιοι και για, το, ε, για, τις ΜΑΝ ε, και όλες τις ε, εξαρτώμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο περιοχές. Αυτά λοιπόν κάνουμε οι στόχοι μας και το καθεστώς μας υπάρχουν στο καταστατικό μας. Ε, εμείς είμαστε υπόλογοι απέναντι στο Συμβούλιο Υπουργών ε, για θέματα πρόοδου. Τώρα, θα μιλήσω λιγάκι για ε, δικά μας βρήματα στον τρίτο γύρο των αξιολογήσεων. Αυτή τη στιγμή είμαστε ο μόνος οργανισμός που μπορεί να περάσει ένα τέταρτο γύρο μετά από τις συστάσεις που προέκυψαν κατά τον τρίτο γύρο. Ο τρίτος λοιπόν γύρος ε, μας έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να δω συγκεκριμένα την οριζόντια αναθεώρηση την οποία και δημοσιεύσαμε πέρυσι. Τα ευρήματα που θα σας δείξω έχουν σχέση με τις ε, χώρες Μάνεβαλ, αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι εξίσου σημαντικά και για άλλες ευρωπαϊκές νομολογίες ε, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη και την υποχρέωσή μας για πρόληψη. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος και αυτό ε, είναι εντυπωσιακό κυρίως όσον αφορά την πρόληψη ε, με την οποία λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Γνωρίζουμε ότι πολλά χρήματα δαπανώνται για πρόληψη από τον ιδιωτικό τομέα. Βλέπετε λοιπόν ότι όλες οι χώρες της Μανιβάλ ε, έχουν ασχοληθεί με την προληπτική νομοθεσία. Αυτή έχει ενισχυθεί καθώς ε, προκύπτουν και συγκεκριμένες ε, προδιαγραφές που να αφορούν στον εντοπισμό και στην επαλήθευση των αποδεκτών ε, στις χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σε σχέση με την οδηγία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την τρίτη οδηγία. Υπάρχουν και πολύ καλά ε, αποτελέσματα όσον αφορά στην υποχρέωση για τήρηση στοιχείων. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί, Γιατί είναι απαραίτητο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να κρατάνε σωστά στοιχεία για τις σχέσεις τους με τους πελάτες έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ανατρέξει στις συνδιαλλαγές 66% των ε, κρατών ε, τήρησαν τις υποχρεώσεις τους. Στον τραπεζικό και στον οικονομικό τομέα η συμμόρφωση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλους τομείς ε, και ιδιαίτερα προβληματικά είναι τα όσοι ασχολούνται με, την, με το συνάλλαγμα η εποπτεία βεβαίως και είναι μεγαλύτερη στον χρηματοψηφιακό τομέα και ενώπιον του κυρίου Ραφαέλ μπορώ να πω ότι υπάρχουν επαγγελματίες και λιγότεροι επαγγελματίες που ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα. Οι τράπεζες και οι μεγάλοι χρηματοψηφιακοί οργανισμοί είναι οι μεγαλύτεροι ε, θεσμοί που αναφέρονται για τα θέματα που μας απασχολούν. Και βεβαίως ε, πρέπει να πω ότι οι δικηγόροι συνήθως δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες. Το ίδιο ισχύει και για άλλους ε, μη ε, οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Θα ήθελα τώρα, ακριβώς ε, λόγω των πόρων που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας στο, στην πρόληψη, θα ήθελα όλα αυτά να τα συγκρίνω με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου. Και όλα αυτά είναι σημαντικά. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οι ε, καταδίκες, η δίωξη και οι καταδίκες αυξάνονται, αλλά τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι περιορισμένα σε αρκετές χώρες. Έχετε λοιπόν μπροστά σας έναν κατάλογο, ο οποίος ε, καλύπτει την περίοδο από το 2005 έως το 2009, σε σχέση ε, όσον αφορά στις χώρες Μανεβάλ. Αυτός λοιπόν ο πίνακας, επ' αυτού θέλω να πω ότι πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός όσον αφορά τους αριθμούς. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα των αξιολογητών είναι να αποκτήσουν ε, στατιστικά δεδομένα που να βγάζουν νόημα γιατί πολύ συχνά ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και ασυνεπή δεδομένα, ε, με διαφορές, άλλα υποβάλλονται στους ε, υπουργού δικαιοσύνη, άλλα υποβάλλονται στις διοκτικές αρχές. Αυτό λοιπόν ε, που έχει σημασία είναι πώς γίνεται ο χειρισμός αυτών των δεδομένων. Πάντως, σε γενικές γραμμές θέλω να πω ότι οι περισσότερες χώρες Στις περισσότερες χώρες προκύπτει καταδίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αλλά περιορισμένα. Και αν δει κανεί τα συμφέροντα που έχουμε εμεί για την αποτελεσματικότητα, το πόσο μα ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, από εκεί μπορεί κανεί να συνάγει και συμπεράσματα για το πόσο σοβαρή είναι η δίωξη. Εδώ βέβαια η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Η διαφάνεια δείχνει ότι δεν υπάρχει άμετη σχέση ανάμεσα στις, στα εγκλήματα και στα ε, κέρδη που προκύπτουν. Πολλές φορές ρωτάμε ποια είναι αυτά τα δικήματα που ε, αποφέρουν μεγάλο κέρδος. Δώστε μας ένα κατάλογο εμπορία ανθρώπων, παραδείγματος χάρη και άλλα. Και είδαμε τα δικήματα και δεν έχουν αυτά καμία σχέση με τα κέρδη τα οποία πραγματικά προκύπτουν από σοβαρά αντικείμενα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι οι ιδιοκτικές αρχές, ε, και ανήκα και εγώ κάποτε σε αυτές, οι ιδιοκτικές λοιπόν αρχές ε, επιλαμβάνονται των ε, απλών υποθέσεων. Ας πούμε, αν διώκεται κάποιος για απάτη, τελικά αυτό ε, δεν ε, αντικατοπτρίζεται στην ποινή που του επιβάλλεται. Γι' αυτό ε, λοιπόν και προέκυψε το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Αυτό καθεαυτό. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν διώκονται εκείνοι οι οποίοι κάνουν το ξέπλυμα για ε, λογαριασμό κάποιου τρίτου. Αυτές είναι και πιο δύσκολες περιπτώσεις, είναι δύσκολο να αποδειχθούν, αλλά αυτή είναι εκείνη, ας πούμε αυτό μπορεί να είναι δικηγόροι, λογιστές, αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι ξεπλένουν το χρήμα για ομάδες ε, οργανωμένου εγκλήματος, ε, για εγκληματίες που ζουν με πολύ ψηλό ε, lifestyle, τρόπο ζωής. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οι προσπάθειες των αστυνομικών αρχών, διοκτικών αρχών, δεν είναι σε άμεση αναλογία με τις προσπάθειες που καταβάλει ο ιδιωτικός τομέας. Πολύ σύντομα θέλω να πω επειδή πολλοί αναφέρθηκαν σε STRs, ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τα STRs, δηλαδή με αυτές τις εκθέσεις περί υπόπτων, ένα από τα σημαντικά είναι ότι ποτέ ε, δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια καταδίκη που να προκύπτει μέσα από το σύστημα της καταγραφής υπόπτων. Ε, γνωρίζουμε περιπτώσεις όπου αυτά τα, αυτές οι εκθέσεις ε, βοήθησαν την δίωξη, αλλά ε, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Το 50% των κρατών στέλνουν λιγότερο από το 10% αυτών των ε, εκθέσεων που λαμβάνουν περιπόπτων ε, στις αστυνομικές αρχές για περαιτέρω έρευνες. Άρα δηλαδή το ερώτημα τι γίνεται τελικά με αυτές τις εκθέσεις. Και αν τα βάσει κανείς την έκθεση ε, το θέμα δεν είναι πώς χειρίζεται κανείς αυτές τις εκθέσεις αλλά τίθενται ερωτήματα για την ποιότητα και τον αριθμό αυτών των εκθέσεων που λαμβάνουν οι διοκτικές αρχές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν περισσότεροι πόροι που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας. Πρέπει να έχουμε ε, ένα πιο αυστηρό σύστημα κατασχέσεων, ε, το οποίο ε, θα συμβαδίζει με την πρόληψη, το ε, δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στους εγκληματίες με υψηλή ποιότητα ζωής. Ε, υπάρχει και σχετική σύμβαση της Βαρσοβίας. Επίσης ε, πρέπει να βελτιωθεί η διεθνής συνεργασία και αυτό είναι ένα τομέα που τον καλύπτει η συνθήκη της Βαρσοβίας. Είναι σημαντικό κυρίως για όσους ε, είναι αρμόδιοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία για περιπτώσεις ε, όπου ε, δεν υπάρχει δέσμευση με βάση την καταδίκη και αυτή η σύμβαση έχει τις πιο δεσμευτικές διατάξεις καλούνται οι χώρες να συνεργάζονται με άλλες που έχουν τέτοιες μορφές κατασχέσεων. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα κατά τη. Ε, ελπίζω αυτά που είπα να σας βοήθησαν. Ευχαριστούμε κύριε Ρίγκοτ. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να καλωσορίσω και εγώ 28 μαθητές ε, από το Λίκιο του Κορέτζου από την ε, <clears throat> Ρέτζιο Μίλια. Καλώς ήρθατε στις εργασίες μας. Τώρα, πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που έθεσα ήδη σήμερα το πρωί, αλλά δεν να απαντήσεις. Ίσως λοιπόν κάποιος από εσάς τους τρεις να μπορούσε να μου δώσει τουλάχιστον μια πρώτη απάντηση, γιατί ακούσαμε για το ρόλο τραπεζών στο θέμα του ξεπλήματος. Όμως φαίνεται σαν να είναι δορυφορικός ο ρόλος των τραπεζών. Αντίθετα όμως, διαφορετικά πράγματα μας λένε τα δεδομένα, τα γεγονότα, ότι έχουν θεμελιώδη ρόλο, αρνητικό ρόλο οι τράπεζες στις δραστηριότητες του ξεπλήματος και στην πραγματικότητα αυτό που το πληρώνουν είναι οι πολίτες. Εγώ σήμερα το πρωί Έθεσε ένα παράδειγμα στους ε, προηγούμενους ομιλητές και ανέκυψε ένα ζήτημα και μάλιστα είδαμε και κάτι σήμερα το μπορείς στις τελικές εφημερίδες. Ορισμένες μεγάλες ε, τράπεζες και επικεφαλής η έδωσε, έχουν δώσει όλες μαζί, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ με μορφή αμοιβαίων δανείων σε ένα νεαρό 20 χρονών που δεν είχε κανένα εισόδημα, δεν εργαζόταν, γεννήθηκε το 1990 αυτό το παιδί. Του είχαν δώσει ένα εκατομμύριο ευρώ για, ως αμοιβαίο δάνειο για να αγοράσει ένα μεγάλο εστιατόριο χωρίς καμία πληροφορία. Δηλαδή, το παιδί αυτό. Η έρευνα, γιατί κατόπιν η τελική εισαγγελία προφανώ κατήσχησε τα πάντα και φυσικά ακύρωσε την πίστοση. Από την έρευνα πρόκειψε ότι ο υπάλληλο απλώ έγραψε σε ένα κομμάτι χαρτί ότι ο νερό <laughs> ανήκε σε μια καλή οικογένεια. Και καλή οικογένεια τελικά ήταν ε, ε, μαφιόζη. Ε, και ότι ήταν ένα σίγουρο άτομο και μπορούσε να του δώσει αυτή τη τεράστια πίσταση. Τώρα αυτό που ανέκυψε και ποιος ξέρει πόσες υποθέσεις δεν έχουμε δει, δεν έχουν ανακύψει στο φως και ε, αυτό είναι τεράστια ζημία. Ε, Τι είμαι λοιπόν, ποιος έλεγχος υπάρχει και προφανώς ε, υπάρχει ένας αρνητικός ρόλος των τραπεζών στις δραστηριότητες νομιμοποίησης παρανομών εσόδων. Ήθελα να σας πω ότι οι διαδικασίες υπάρχει ε, απουσία ε, μεγάλων υποθέσεων, πολλές φορές εισαγγελία παρακολουθεί τις μικρές υποθέσεις και εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι ε, υπάρχει απουσία καταγγελίας για αυτές τις εκθέσεις, τις STR και εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή Ποιο ξέρει τι βρίσκεται ακόμη στο σκοτάδι. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιακολίνο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Ακούσαμε τις παρεμβάσεις, όμως δυστυχώς έχασα την παρέμβαση της πρώτης εισηγήτριας. Άχουσα βέβαια το, δεύτερο και το τρίτο μιλητή. Σήμερα ακούσαμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για τις δραστηριότητες μας. Η Ευρώπη θέλει μια κοινή γλώσσα για να καταπολεμήσει την ομοιοποίηση παράνομων εσόδων και τη διαφθορά και οι δύο αναφερθήκατε ε, στην νομοθεσία, ότι η πρώτη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρονολογείται το 1986. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση έχει ε, συνάψει και τη συμφωνία πριν κάποιο καιρό για την ανταλλαγή πληροφοριών για την της τρομοκρατίας μέσω SWIFT. Όταν εσείς μιλάτε τώρα για αυτή την κουλτούρα, για αυτόν τον πολιτισμό ε, της καταγγελίας ίσως να μην είναι τόσο ισχυρή αυτή η κουλτούρα, όμως όταν καταλαβαίνουμε εκεί η Ευρώπη τώρα προχωρά με μια νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανοσόδων, για μια νέα οδηγία για τη δίμευση και σίγουρα υπάρχει και η απέτηση στο κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα να έχουμε και μία συμφωνία με τις τρίτες χώρες, γιατί οι αγορές είναι πλέον παγκόσμιες και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Τώρα, από τη δική σας σκοπιά που δραστηριοποιήσετε σε αυτόν τον τομέα, τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο στάδιο ολοκλήρωσης της σύνταξης οδηγίας για την καταπολέμηση τη νομιμπήσης παράνομων εσόδων και της οδηγίας για τη δίμηση. Πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας για να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό το μέτρο της δίμευσης και της κατάσχεσης. Εσείς ε, τι πιστεύετε σε σχέση με τα νομοθετήματα που εξετάζουμε και σε σχέση και με το τελικό φάκελο που θα μας επιτρέψει να προστρέξουμε στις συμφωνίες συνεργασίας που βασίζονται φυσικά στην εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να καταπολεμήσουμε την παραοικονομία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Ο κύριος Νιούτον τάνια για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλήτες. Η κυρία από την τράπεζα πρώτα. Δεν κατάλαβα τι εννοούσατε όταν λέγατε έχουν πρόσβαση οι τράπεζες στα μητρώα των μετόχων. Τι εννοεί αυτό. Και εγώ μπορώ να τα δω. Ίσως να μου το εξηγήσετε γιατί δεν το κατάλαβα. Τον κύριο Ραφαέλ. Πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και πολύπλοκη παρέμβαση. Μιλήσατε για την επίλυση και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το διαμεθοριακό έγκλημα, όχι τα εθνικά. Μόνο το διαμεθοριακό, το διεθνές. Είπατε επίσης πρέπει να πείσουμε την κοινωνία των πολιτών. Τι εννοεί αυτό. Οποιονδήποτε δεν είναι τράπεζα, είμαι και εγώ που κοινωνία των πολιτών. Ποιος είναι, ποιος δεν είναι με την εμπειρία που έχετε ίσως να μας τα εξηγήσετε. Επόμενο, είπατε ότι υπάρχουν πολύ μικρά ποσά που μεταφέρονται από μικρά γραφεία. Αυτά έχουν γίνει ποτέ αντικείμενο πλησίματος βρωμίκου χρήματος. Τέλος, με την πεντηκονταετή σας εμπειρία, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να συστήσουμε και εμείς οι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας. Τι μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα και προς τον τελευταίο που ήταν επίσης πολύπλοκη η ομιλία του και μιλούσε και πολύ γρήγορα. Ελπίζω να μας τη δώσετε και γραπτός μετά, αλλά είπατε πολλές φορές, μιλήσατε για τη συνθήκη της Βαρσοβίας. Εδώ με το η Πάντ μου είδα στο Google ότι αφορά τους ε, επιβάτες αεροπορικών εταιριών την ίδια συνθήκη εννοείται και εσείς. Άλλοι δεν μάλλον, δεν όχι την ίδια. Τι Βαρσοβία είναι αυτό. Αυτό όλο στο Google. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Θα δώσουμε και πάλι το λόγο στην ε, κυρία Σίμπερο και κατόπιν ε, κυρία Ράφαελ και Το έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Απαντήσω πρώτα σε εσά. Μιλήσατε για μια συγκεκριμένη υπόθεση σε ένα συγκεκριμένο κράτος που το χειρίστηκε χρήστηκαν συγκεκριμένες αρχές. Δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοια πράγματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν στους εσωτερικούς μηχανισμούς. Όπως σας είπα και τεχνολογικά και ανθρώπινα δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια πράγματα ή ατυχήματα ή συμβάντα. Μία ευρωπαϊκή νομοθεσία εναρμονισμένη χρειάζεται για να μην επιτρέπονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Τώρα για τα ερωτήματα του κυρίου Νεύτων Ντάν. για τα μητρώα πρώτον. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να γνωρίζουν τη δομή και την ιδιοκτησία των πελατών και πελατησών τους. Μερικά έχουν μητρώα όπου εμφαίνονται όλα αυτά, τι μετοχές έχουν κλπ. Αλλά δεν συμβαίνει σε όλα τα κράτη και ούτε είναι υποχρεωτικό ακόμα στο επιχειρησιακό δίκαιο ή στο δίκαιο των επιχειρήσεων. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να τηρούν εμπορικά μητρώα που μπορεί να εμφαίνονται και από τον Google αλλά δεν υπάρχει κανένα νενομισμένο μητρό ενημερωμένο για όλα τα κράτη-μέλη. Το ζητάμε αυτό, το ζητάμε, το ζητάμε. Να έχουμε τουλάχιστον πρόσβαση σε σαφή και ενημερωμένη ενημέρωση, πληροφόρηση. Ενημερωμένη πληροφόρηση, πληροφόρηση. Αυτά. Αυτά. Um, Μάλιστα, με βάλατε κάτω από το φως του προβολέα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας ε, παρουσιάσω την εμπειρία 25 χρόνων μέσα σε 5 λεπτά. 50. Η κοινωνία των πολιτών στην οποία αναφέρθηκα θα πρέπει να περιοριστεί στο ρυθμισμένο τομέα, δηλαδή στο τομέα που είναι ρυθμισμένο τώρα από διαδοχικέ οδηγίε και έχουν ε, μεταφερθεί στο ιστορικό δίκαιο. Όμως ε, Μιλάμε για ένα μεγάλο κύμα το κοινωνία των πολιτών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχείτε για ανθρώπους ε, ε, οι οποίοι δεν είναι υπορρύθμιση, ε, μιλώ για αυτούς που σέβονται το νόμο και έχουν υποχρέωση στον νόμο να επαγρυπνούν προκειμένου να υποβάλουν σε εκθέσεις. Και κάτι που θέλω να πω για την υποβολή εκθέσεων. Δεν ξέρω αν μπορεί να μεταφραστεί σε νομοθεσία ή σε Υπάρχει μία εντύπωση ότι αν είναι επίγουσα μία συλλογή και πολλές φορές είναι στον ε, χρηματοοικονομικό κόσμο, πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν ε, να στείλουν ε, χρήματα για προσωπικούς ή εμπορικούς λόγους, αρκεί να αναφέρει κάποιος την υποψία του μετά τη συναλλαγή, γιατί ε, φοβάται ότι αν ε, βάλει αυτή την κατοικία και δει ε, ότι υπάρχει συνένεση από τη μονάδα χρηματικών πληροφοριών, ε, τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη συναλλαγή και από μια απόκριβη σκοπιά και θα μου πει και συνάδελφος εδώ εκ δεξιών, αν κάνω λάθος, οι μεγάλες τράπεζε λιανικών υπηρεσιών ε, πρέπει να κάνουν μια κρίση πολύ γρήγορα για το αν χρειάζεται ε, τη συνένωση πριν τη συναλλαγή ή αν αρκεί αυτές ε, να κάνουν μια γρήγορη αναφορά από μια σκοπιά πληροφοριών και να κάνουν τη συναλλαγή χωρίς τη συνένεση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα. Και να πω και κάτι ακόμη. Είπατε για κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί. Είναι κάτι που, για το οποίο δεν έχετε πολύ μεγάλη επιρροή μάλλον. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταρχήν, το οικονομικό έγκλημα, μιλάμε και για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, δεν είναι στην, στον κατάλογο προτεραιοτήτων των περισσότερων διοκτικών αρχών των αστυνομικών δυνάμεων. Είναι πολύ κάτω στον κατάλογο και αν προσθεθεί σαν αδίκημα σε κάποια δίκη, αυτό γίνεται για κοινικού λόγους, ε, είτε για να τιμωρηθεί κάποιο με υψηλότερη ποινή, ή για να υπάρχει πιο εύκολα μία απόφαση περιδίμευσης. Όμως ε, δεν δίνεται προτεραιότητα στην καταπλώμηση του οικονομικού κλίματος. Ε, τώρα τα γραφεία αποστολής χρημάτων. Κάνατε μια αποφαση περιδίμευση. ομως δεν δινεται προτεραιοτητα στην χρήσιμη αποστολή χρηματων κανατε μια πολυ χρησιμη ερωτηση και χαίρομαι που την απαντήσατε εσεί, γιατί αν την απαντούσα εγώ θα με κατηγορούσατε ότι είμαι παρτιζάνος. Η απάντηση είναι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία για το που ε, βρίσκεται κυρίως η ζημία. Δεν ξέρουμε αν αυτά είναι περισσότερο μεγάλες τράπεζες ή κάποια άλλα γραφεία αποστολής χρημάτων, γιατί προφανώς οι διοκτικές αρχές φοβούνται ότι αυτά τα γραφεία που στέλνουν σχετικά μικρά ποσά, συνήθως από 50 μέχρι 500 λίρες, ε, θα κάνουν smurfing, δηλαδή θα σπάνε τα χρήματα σε μικρές δόσεις. Και αυτό είναι ένας φόβος, αλλά δεν έχουμε κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Είναι απλώ ένα φόβος που έχει εκφραστεί από τη ΣΟΚΑ και από άλλες διοκτικέ αρχές. Αλλά δεν υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξέρω ότι σχεδόν ε, κατανάλωσα και τα πέντε λεπτά για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό θα ήταν είναι πολύ περίεργο κάποιος νομικός να το πει αυτό σε εσά, αλλά αν ε, έχουμε τόσο λίγες διώξεις, θυμηθείτε, στο Ηνωμένο Βασίλειο φτάσαμε πολύ κοντά στο να αποποινικοποιήσουμε ε, τους ε, κανονισμούς ε, περί νομοποίησης εισόδων. Υπήρξε συζήτηση στο και γιατί κάποιοι άνθρωποι που ασκούν επιρροή περισσότερο από μένα ε, είπαν σας παρακαλούμε μην ε, τους γιατί ακόμη και αν δεν υπάρχουν δείξεις τότε ουσιαστικά ε, θα υποβαθμίσετε και την αξία της τήρησης αρχείων αλλά υπάρχει πάντα ξέρετε αυτή η ένταση Δηλαδή, συνεχώς ε, μιλάμε για το άχθος ε, της ρύθμισης ε, και πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα εγώ να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο τελευταίος ομιλητής, δηλαδή το να γίνει, να ποινικοποιούμε τις κανονισμούς περί ξέπλυμα βρώμικους χρήματος. Αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν υπάρχουν ποινικέ κυρώσεις οι διεθνείς ε, προδιαγραφές ε, ε, προβλέπουν είτε ποινικέ είτε διοικητικέ κυρώσεις σε αυτούς τους προληπτικούς οργανισμούς. Άρα δηλαδή ποινικοποίηση είναι κάτι που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης πριν πάω στη σύμβασή μας θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άλλα πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν σχετικά με τα γραφεία συναλλάγματο ε, και αυτού ε, που προωθούν το χρήμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις ε, δίωξης από ό,τι θυμάμαι όπου μεγάλα γραφεία συναλλάγματος στο Λονδίνο αποκαλύφθηκε ότι ήταν η βιτρίνα του ξεπλήματος ε, και ε, γι' αυτό το λόγο εκδόθηκαν και εντολές ε, κατάσχεσης για σημαντικά ποσά. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε το ρόλο των γραφείων συναλλάγματος, ανταλλαγής συναλλάγματος. Στον τομέα αυτό, σε πάρα πολλές χώρες, ε, έχουμε πάρα πολλούς που εμπλέκονται σε αυτά τα γραφεία ε, που στέλνουν τα χρήματα. Ε, βεβαίως, δεν ξέρουν τόσο καλά τους κανονισμούς και πολλές τράπεζες εδώ στις Βρυξέλλες, ακόμα και στο Λονδίνο, Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει να ευαισθητοποιηθούν ε, σε αυτούς τους τομείς οι αρμόδιοι για, τις, για τους κανονισμούς που ισχύουν. Υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά ε, την σύμβαση της Βαρσοβίας, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τίτλο. Είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για, την, ε, για το ξέπλυμα χρήματος, για την κατάσχεση ε, των αποτελεσμάτων εγκλήματος ε, και τρομοκρατίας. Ο λόγος λοιπόν που σας τα λέω αυτά είναι όχι γιατί πρόκειται για σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά διότι έχουν σχέση με αυτά που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή το έγκλημα δεν τελειώνει στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, ε, οργανωμένες ε, ομάδες εγκλήματος μετακινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, γύρω-γύρω από την Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη και το καθεξής. Πρόκειται δηλαδή για μια πολύ διεθνοποιημένη μορφή εγκλήματος. Είναι απαραίτητο να υπάρχει καλή ε, νομική αρρωγή ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες, εντός και εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι όταν κάνετε την ερώτηση είπατε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν ρυθμίσεις, κανόνες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ακριβώς αυτό δεν θέλουμε να υπάρχει, δηλαδή διμερείς ε, ε, ρυθμίσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα εργαλείο να αφορά περισσότερα κράτη και όσοι προσυπογράφουν μία συμφωνία να γνωρίζουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας είπα, και ίσως τα είπα πολύ γρήγορα στην εξήγηση, το συγγνώμη γι' αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι χώρες ε, εφαρμόζουν το πρωτόκολλο ε, και τη σύμβαση για την αμοιβαία νομική συνδρομή, τότε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε, λέω σκόπα θα έπρεπε και όχι μπορούν, θα έπρεπε να προσφέρουν ε, πληροφορίες για το κατά πόσον κάποιος έχει τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη χώρα, να δίνουν το ιστορικό ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, δεν υπάρχουν κάποιες ρήτρε προστασίες, και επίσης ε, να ε, επιτρέπουν και τον μελλοντικό έλεγχο αυτού του τροπεζικού λογαριασμού να ζητάνε από την τράπεζα να παρακολουθεί το λογαριασμό κάποιου υποπτού βέβαια και πάλι κάτω από συγκεκριμένους όρους που προβλέπονται. Εντάξει, αν αυτά γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώ. Αν όμω χρειάζεται κανεί πληροφορίε από τη Ρωσία ή από την Ουκρανία ή από τι χώρε Μάνεβαλ στα Βαλκάνια, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία επικύρωσε τη σύμβαση και η Αλβανία αρκετές χώρες, οι μεγάλες χώρες ε, θα την ε, επικυρώσουν σύντομα. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχουν και αυτές επικυρώσει θα ζητήσουν το ίδιο πράγμα από την Ουκρανία όπως και από τη Γαλλία και την Αλβανία. Αυτό σημαίνει διεθνή συνεργασία, κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και η κατάσταση είναι η εξή. Έχουμε 13 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν συμπεριλάβουμε και την Κροατία, που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση. 10 και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, μονογράψει αλλά όχι επικυρώσει ακόμα τη σύμβαση και σε πάρα πολλά ε, βήματα που καλούμεθα ασκούμε πίεση στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνουν όλα τα κράτη και επειδή αυτή η ερώτηση τέθη από το Ηνωμένο Βασίλειο, με συγχωρείτε, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο ούτε έχει υπογράψει, ούτε έχει επικυρώσει ακόμα τη σύμβαση. Και έγιναν ε, ερωτήσεις ε, στο, στη Βουλή των Λόρδων. Εγώ έδωσα κάποια στοιχεία και μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προεδρεύσει στην Επιτροπή Σύνταξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι λοιπόν σημαντική αυτή η σύμβαση και είναι σημαντικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθεί μεγαλύτερη σημασία ε, στα εργαλεία που υπάρχουν και να προσπαθεί κανείς να τα επεκτείνει και πέρα από την Ευρώπη για να υπάρχει καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας για τις παρεμβάσεις τους. Σας καλώ, όπως έκανα και με τους προηγούμενους καλεσμένους μας, να αφήσετε την τεκμηρίωσή σας στη γραμματεία και να μας στείλετε γραπτό στη σκέψη σας, αν το θεωρείτε σκόπιμα. Τώρα θα καλέσω τους επόμενους ομιλητές να έρθουν εδώ στο βήμα. Πριν όμως να κάνω μια ανακοίνωση. Ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους και οποιονδήποτε το επιθυμεί να συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα στην προβολή της ταινίας. Ε, ε, ο δεύτερος καιρός ε, και αναφέρεται εκεί στο μικελιό που έγινε στην Οδόντα Μέλιο θα γίνει η ε, προβολή στην αίθουσα ASP 1G3 και θα είναι η κυρία και θα είναι και ο Γενικός Εισαγγελέας Καρτινάτο και ο Χάνης Βόμποντα. Τώρα, περνάμε στο τέταρτο κλάστερ, έλεγχο των χρηματοοικονομικών όρων πώς αντιμετωπίζουμε περιοχές που δεν συνεργάζονται και πώς ελέγχουμε τις ταμιακές ροές από και προς την Ευρώπη. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Φίντλερ από τη Γερμανική Αστυνομία που θα σας μιλήσει για την εμπειρία της ε, Γερμανίας ε, για την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων σε σχέση με τις ε, περιφέρειες, με τις περιοχές που δεν συνεργάζονται. Επίση τον κύριο Κάρβερ που θα μας μιλήσει για το ρόλο των επαρχιών ε, που δεν συνεργάζονται στο ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματο και επίση τον κύριο Κάρλο Βαν Χελίνκομ από την Γερόπολη που θα μας μιλήσει για την επιχείρηση Αθηνά και για τα μέτρα για την αποτροπή των ταμιακών ροών ως στοιχείο για την αποτροπή του ξεπλήματος Βρώμικου χρήματος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φίτλερ που θα μας μιλήσει για τη γερμανική εμπειρία στην εφαρμογή του νόμου, στις έρευνες ε, για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος σε σχέση με τα μη συνεργαζόμενα εδάφη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση. Και για μας είναι μεγάλη τιμή ε, το ότι μας δίνεται η ευκαιρία να σας μιλήσουμε για τι συμβαίνει στην πρακτική. Εγώ μιλάω για την επαγγελματική οργάνωση των ε, Γερμανών ε, υπαλλήλων δίωξη του εγκλήματος. Εγώ ε, ασχολούμαι αρκετό καιρό με το οικονομικό έγκλημα και εδώ και 1,5 χρόνο ασχολούμαι κυρίως ε, με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ε, και με όλα τα προβλήματα που έχουμε στη Γερμανία. Βεβαίως η επικεφαλίδα της ομιλίας μου είναι πάρα πολύ ευρεία και προσπάθησα να την χωρίσω σε τμήματα Θα ήθελα να δούμε λιγάκι τον όρο έλεγχος, κατά πόσον αιτιολογείται αυτός ο όρος ή όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω, καταρχήν αφορά την πρακτική εμπειρία. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς συναδέλφους πριν έρθω εδώ για να σας ε, αναφέρω και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, ε, στο πρώτο κομμάτι της ομιλίας μου ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε επιλεγμένους χώρους, σκιώδεις, γκρι χώρους που μας δημιουργούν πολλά προβλήματα στις ανακρίσεις μας. Στο δεύτερο τμήμα θα μιλήσω λιγάκι για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της Γερμανίας, δηλαδή τι συμβαίνει όταν άλλες χώρες απευθύνονται σε εμά για δραστηριότητες της ε, ε, ξεπλήματος ε, και επιθυμούν να υπάρξει δέσμευση στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων. βεβαίως, επειδή το θέμα είναι και επίκαιρο, ίσως θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το ξέπλυμα χρήματος σε μια χώρα. Αυτά βέβαια σχετίζονται με αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Και στο τελευταίο τμήμα της ομιλίας μου θα ήθελα να καταθέσω επικοδομητικές προτάσεις. Λοιπόν, στην αρχή είχα πει ότι έχουμε γκρι φεούς χώρους οικονομικών συναλλαγών. Η εμπειρία την οποία έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, κατ' ουσίαν, είναι εμπειρία εκείνη ε, που υπάρχει και σε άλλες χώρες. Ένα από τα κράτη με τα οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό είναι κοντά μας είναι η Κύπρος. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές ε, ανακρίσεις ε, που καταλήγουν εκεί, στην Κύπρο. Και αυτό οφείλεται στο ότι εκεί ε, ιδρύονται εταιρείες ψεύτικες, απλώς εταιρείες οι οποίες έχουν κατ' ουσίαν ε, εταιρείε φάντασμα. Αυτό λοιπόν αφορά κυρίως και μας ε, ενδιαφέρει όταν επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε τις ε, ροές του χρήματος. Η νομική βοήθεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για σκεφτείτε το να θέλει κανείς ε, να επιταχύνει μια διαδικασία ε, στον βαθμό που δεν τα καταφέρνει επηρεάζεται και η διάρκεια της, ε, της σύλληψης, της φυλάκισης. Οι προϋποθέσεις από την Κύπρο προς εμάς και οι όροι που υποβάλλονται είναι ε, πάρα πολύ αυστηροί, ε, δηλαδή δεν αρκεί απλώ να τους δώσουμε του λογαριασμού, αλλά μας ζητούν να τους πούμε συγκεκριμένα ποιον ακριβώς δρόμο ακολούθησαν, ποια πορεία ακολούθησαν ε, τα αντικείμενα αυτά. Κατόπιν υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι πολύ επίκαιρες και έτσι λοιπόν ε, μπορούμε να ρίξουμε ε, μια ματιά στην δυσκολία των ε, ανακρίσεων. Έχουμε μια επίκαιρη περίπτωση όπου έχουμε ένα πλοίο στο Κουρασάο το οποίο είναι καταχωρημένο σε νεολόγιο των νήσων της Μάνχης και η εταιρεία Φάντασμα έχει την έδρα της ε, στο, Γιβραλτά, στο Γιβραλτάρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ε, χρονοβόρα είναι η διαδικασία. Και έτσι δεν είναι απλό να αποκαλύψει κανείς ε, περιπτώσεις όπου το θέμα δεν είναι να έρθει κανείς σε επαφή με τους ανακριτές, αλλά τις, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα τα οποία εξάγει να τα εντάξει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κόνγκ. Και ε, παρουσιάζουν αυτές οι δύο πόλεις σε μεγάλο ενδιαφέρον για τους εγκληματίες. Ε, ε, και αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η Γερμανία είναι πολύ κοντά στην Ελβετία, άρα δηλαδή είναι αυτό αποτρεπτικό. Ε, στην Ελβετία παρόλα αυτά συγκεντρώνεται περίπου το 30% όλων των περιουσιακών ε, στοιχείων που προκύπτουν από τέτοιες ε, παράνομες ενέργειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε λιγάκι την εικόνα. Αφενός έχουμε την συγκεκριμένη συνεργασία με τις εισαγγελίε, με τους συναδέλφους των αστυνομικών αρχών. Το πρόβλημα με την νομική αργή αρρωγή είναι η διάρκεια. Ε, πολλές φορές, ε, σας είπα, είναι πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ρήτρε προστασίας. Οι ε, ύποπτοι και οι εναγόμενοι μπορούν να καταθέσουν εφέσεις και διαμαρτυρίες, καταγγελίες, άρα δηλαδή δεν είναι εύκολο να αποκαλύψουμε συγκαλυμμένες και κλειστούς λογαριασμούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, όπως ε, σας είπα, οι εταιρείε ε, φάντασμα που συνεργάζονται με άλλες εταιρείε. Αυτό είναι τόσο καταστροφικό που παραδείγματο χάρη σε πολλές φορές ε, παρατηρούμε ότι οι σε μια εταιρεία ε, είναι οι ίδιοι οι οποίοι έχουν συστήσει μια εταιρεία φάντασμα. Ε, βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες μας. Και όσον αφορά τις ε, τράπεζες, επειδή ετέθη αυτό το θέμα, πρέπει να πούμε ότι η εμπειρία μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Αφενός είναι αλήθεια ότι και στη Γερμανία φτάνει το πάνω από 90% όλων αυτών των ε, παράνομων ε, ε, δραστηριοτήτων. Από την άλλη όμως έχουμε και μεγάλες υποθέσεις στην Ελβετία. Η UBS είναι μια περίπτωση που βγήκε στον τύπο και άλλο ένα ίδρυμα στην Ελβετία το οποίο είχε καλύψει ένα δις ευρώ και τελικά γλίτωσε με μία ποινή μόνο 300.000 ευρώ. Άρα δηλαδή ε, καταλαβαίνετε ότι εμείς θα επιθυμούσαμε αυστηρότερες ποινές γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί ένα τέτοιο χρηματοψωτικό ίδρυμα ε, παράνομο που ασκεί παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να δύναται να συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην Γερμανία. Αλλάζω τώρα λιγάκι ε, την εικόνα που θέλω να σας παρουσιάσω και σε εμά συμβαίνουν πολλά από αυτά που συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Η νομική αρρωγή κατά την άποψή μου είναι ένα από τα κλειδιά για να σημειώσουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει μία περίπτωση επίκαιρη αρκετά επίκαιρη ενός Ολλανδού ε, εμπόρου ναρκωτικών ε, ο οποίος είχε ένα τεράστιο ποσό ως ε, κέρδος του από το λατρεμπόριο ναρκωτικών. Αγόρασε ε, ακίνητη περιουσία στη Γερμανία, είχε και χρήματα στους ε, τραπεζικούς λογαριασμούς. Βέβαια εμείς ε, θελήσαμε να δούμε πού ακριβώς ε, απέκτησε ακίνητα στη Γερμανία. Επειδή όμως όλο αυτό ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρο και δεν μπορούσαμε και να το τεκμηριώσουμε απόλυτα, τελικά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δεν μπορέσαμε να του κατάσχουμε ούτε ένα σεντ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ε, πόσο σημαντικό είναι να δει κανεί ε, την αποτελεσματικότητα. Καλό να υπάρχουν πολλοί κανονισμοί, αλλά να υπάρχει και αποτελεσματικότητα, γιατί αυτό είναι το δικό μας το καθημερινό πρόβλημα. Αυτό αφορά και το, την απόφαση πλαίσιο για την ε, διασφάλιση και την προστασία. Ε, οι απαντήσεις δίδονται με διαφορετικό τρόπο, ακόμα και αν υπάρχει η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή αυτή εφαρμόζεται διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν χώρες όπου απαιτείται ε, τα τοπικά δικαστήρια να αποκτήσουν απόφαση από εθνικό δικαστήριο. Βεβαίως ήταν σκόπιμο να υπάρχει απόφαση μιας άλλης χώρας που να τίθεται σε λειτουργία άμεσα ακριβώς όπως συμβαίνει και με το Ευρωπαϊκό Εντάλμα Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ε, το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία. Εδώ πολλά είναι ίδια με αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, ε, με τα ερωτήματα που ε, ετέθησαν, τουλάχιστον όσον αφορά την ευαισθητοποίηση. Σας είπα ότι πάνω από 90% έρχονται των καταγγελιών αφορούν τον χρηματοψηφιακό τομέα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μόνο 20% αφορούν καταγγελίες από, σε άλλους τομείς. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο καταρχήν να υπάρξει ευαισθητοποίηση των άμεσα ενδιαφερόμενων, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όσοι θίγονται από το ξέπλυμα χρήματος επειδή συμμετέχουν στην οικονομική ζωή ε, γνωρίζουν γιατί είναι σημαντικό να καταγγείλουν το ξέπλυμα. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι πολιτικό καθήκον ε, και εδώ ε, η μεγαλύτερη δυσκολία στην όλη συζήτηση. Δηλαδή σε ε, θέματα κρατών και εθνικής ε, πολιτικής ε, ε, το, η ασφάλεια και το αίσθημα της ασφάλειας να προβληθεί. Αυτό όμως αντιμετωπίζει πολλές αντιφάσεις γιατί αν ακούσουμε και αν δούμε τι είδους υποθέσεις μας απασχολούν δεν πρέπει τις υποθέσεις αυτές να τις υποτιμούμε. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό να έχουμε τη βοήθεια των ε, οικονομικών παραγόντων μιας χώρας. Ε, πρέπει να γίνει κατανοητό Ας πάρουμε ένα τυχαίο παράδειγμα, γιατί είναι σημαντικό ένας έμπορος αυτοκινήτων να ξέρει ότι μπορεί να πάρει 70.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο που όμως να πρέπει να το καταγγείλει αυτό στην αστυνομία. Πολλές φορές δεν το ξέρει και δεν το κάνει. Στα ακίνητα το ίδιο. Πριν από λίγο καιρό δημοσιεύσαμε μία μελέτη και αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και παραδείγματο χάρη, όταν μιλάμε για εξαναγκαστικούς πληστηριασμούς στη Γερμανία, είναι δύσκολο ε, να διαπιστώσει κανείς ε, αυτοί που αγοράζουν, που βρίσκουν ε, τα χρήματα, γιατί μπορούν να πληρώσουν με τριτής. Και δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει υποχρεωτικά ισχύει το πόθεν έσχες του αγοραστή. Αυτό δείχνει λοιπόν η μελέτη και καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση. Τέλος, Θέλω να σας πω ότι δεν αρκεί και να υπάρχει μόνο ευιστοποίηση, καλή και αυτή, αλλά δεν φτάνει. Ε, πρέπει να υπάρχει και ε, επανεξέταση, έλεγχος ε, στις τράπεζες, γενικότερα στην οικονομία, compliance, η περίφημη συμμόρφωση. Εμφανίζεται μόνο εφόσον κάτι γίνεται ή εφόσον ασκείται πίεση. Εκεί γίνονται προτάσεις για αυτορύθμιση. Έχουμε λοιπόν εποπτικές αρχές ε, μετά από πολλές ε, διαδικασίες ε, καταγγελιών επί παραλήψη. Έχουμε τώρα πολλές τέτοιου είδους αρχές αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για άμεση αποτελεσματικότητα γιατί έχουμε πάνω από 200 εποπτικές αρχές σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Υπουργείου, παντού. Άρα δηλαδή αν δεν έχουμε εμπειρογνώμονες, αρκετούς εμπειρογνώμονες τελικά δεν θα σημειώσουμε επιτυχία. Και έτσι φτάνω στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας μου και στις προτάσεις ε, που είναι σημαντικές. Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα που πρέπει να εντάξουμε στην πολιτική συζήτηση είναι το μήνυμα ε, ότι η ε, αντιμετώπιση του εγκλήματος είναι πιο φτηνή από το να ασχοληθεί κανείς με τους πόρους, με τα κέρδη που ε, προσπορίζεται η εγκληματικότητα. Η πολιτικοί ε, προφανώς θα πρέπει να θέσουν προτεραιότητες εάν εμφανιστούν περισσότερα φαινόμενα. Σε εμάς ας πούμε στη Γερμανία έχουμε τους ρόκερς, ε, έχουμε τους σαλαφιστές, έχουμε πολλές ομάδες που μας δημιουργούν ε, προβλήματα και σε αυτούς διοχετεύονται οι πόροι και όχι αλλού. Αυτό όμως, γι' αυτό σας είπα, είναι πολύ πιο δαπανηρό το να ασχοληθεί κανείς με τα χρήματα του εγκλήματο και όχι με το έγκλημα το ίδιο. Μπορεί να συγχύει αυτό συνδικαλιστικό, αλλά δεν είναι έτσι. Και επίση, τελικά δεν πρόκειται για την ποσότητα, πρόκειται για την ποιότητα. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση ε, για τις... Ε, τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι ειδικοί, τόσο οι του τμήματος δίωξης εγκληματικότητας όσο και των αστυνομικών αρχών. Και τέλος, ε, τελευταίο κομμάτι και έτσι κλείνω, θα ήθελα να προτείνω το εξής. Σε πάρα πολλούς τομείς δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πολλά. Σε πολλούς τομείς απλά ε, καταλήγουμε σε παραδοχές. Ε, κατά την άποψή μας όμως είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε τις γκρίζες ζώνες για να μπορέσουμε εκεί να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Τζέρεμι Κάρβερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και την Επιτροπή σας για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ την Transparency International Εκπροσωπώ την κοινωνία των πολιτών, γιατί έτσι είχε, κάτι τέτοιο είχε ρωτήσει ο κύριος Νεύτον Ντάν προς τον κύριο Ραφαήλ. Λοιπόν, η Transparency International είναι τώρα αρκετά γνωστή ώστε να μην χρειάζεται να την παρουσιάσω διαμακρού. Εδώ όμως δεν ήρθα για να σας μιλήσω κυρίως για τη διαφθορά, γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε για τη διαφθορά ως πτυχή του ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος. Το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος πρέπει να σταματήσει για να μην μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτά τα παράνομα χρήματα για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή για διαφθορά και οτιδήποτε άλλο. Αν δούμε τους αριθμούς βλέπουμε ότι τα κέρδη από τη διαφθορά διεθνώς είναι 20 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Και μέσω του διεθνούς πιστοτικού συστήματος 1,5 με 1,8 3 εκατομμύρια. Αυτό το σημαίνει ότι αν μπορέσουμε να μειώσουμε έστω και για μόνο 10% αυτή την πληγή θα κάνουμε κάτι σημαντικό υπέρ της κοινωνίας και θα διορθώσουμε σε μεγάλο βαθμό ένα, αυτό το πρόβλημα. Και αυτό χρειάζεται γιατί όλα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ροές αυτές αυξάνονται γεωμετρικά, δεν μειώνονται. Πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί. Επίσης θέλω να αποσαφηνίσω ότι αν και προβλέπετε να μιλήσω για το ρόλο των, των μη συνεργαζομένων περιφερειών στο ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος και υπάρχει πλήρης κατάλογος των περιφερειών και χωρών αυτών όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, η Βολιβία, η Κούβα και ο Ισημερινός. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα χωρίς να μειώνω βέβαια τη σημασία που έχει ο ρόλος των χωρών αυτών ότι οι χώρες αυτές δηλαδή συνεχίζουν να υπάρχουν γιατί χρησιμοποιώντας τέτοια κεφάλαια γιατί δεν μπορούν να βρουν τον τρόπο να ελέγξουν την ροή των χρημάτων από το έγκλημα. Γι' αυτό είναι σημαντικό για αυτές, αλλά όχι για σας ως Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι αυτό το θέμα σας. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στο θέμα των φορολογικών παραδείσων, που είναι γνωστό ότι ε, κάνουν ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος. Το Βανουάτο ας πούμε ή περίεργες νομοθεσίες στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό μικρών χωρών που λειτουργούν ως φορολογική παράδειση. Υπάρχουν και μέλη της Ένωσης. Ορισμένες βρετανικές κτίσεις, 14, που τους έχουν αναφέρει και άλλοι, η Ολλανδία και γαλλικές υπερπόντιες κτήσεις. Όλες αυτές παίζουν κάποιο ρόλο. Αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στους σημαντικότερους από αυτούς τους παραδείσους. Είχαμε πει και πριν ότι η Ελβετία είναι μάλλον ίσως και τμήμα της Γερμανίας. E και πρέπει να σας πω ότι ο σημαντικότερος στην Ένωση είναι το ΙΤΑΒΙΤΑ. Το έχει πει πολλές φορές η Εύα Ζολή όταν ήταν δικαστικός ή ο Γιάννης Μόσκο που πολλές φορές είπε ότι το City του Λονδίνου είναι το μεγαλύτερο πλυντήριο χρημάτων στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια αλήθεια σε όλα αυτά γιατί παράλληλα είναι το μεγαλύτερο πιστοτικό κέντρο του κόσμου. Με συγχωρείτε αλλά Αν είναι δυνατόν, θα ήθελα εσείς να σταθείτε σε αυτή την πτυχή. Μην το θεωρείτε ότι είναι κάτι δεδομένο, να το υπογραμμίσετε. Καλά. Το City του Λονδίνου είναι το μεγαλύτερο χρηματοπλυντήριο του κόσμου. Γιατί έχει τον μεγαλύτερο, τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών. Και δεν χρειάζεται νομίζω να λέμε ότι Υπάρχει μεν το City του Λονδίνου αλλά δεν με εμείς. Το σύστημα είναι σύστημα. Όταν κάνω συζητήσεις στην Transparency International που να προσέξουμε, τι να προσέξουμε, είναι σαφές ότι καλά λέγαμε ότι από τη μία πλευρά της διαφθοράς υπάρχει κάποιος που δωροδοκεί και από την άλλη κάποιος που παίρνει το δώρο. Είναι διπλή σχέση, αμφίδρομη αλλά για τη διαφθορά και οτιδήποτε άλλο συζητάμε εδώ μέσα, τρία είναι τα συμβαλόμενα μέρη. Στη μέση είναι η ενδιάμεση, γι' αυτό είναι στη μέση. Οι οποίοι δεν είναι απαραίτητος διεφθαρμένοι, όσο θέλουν μόνο. Μπορούν να λειτουργήσουν το σύστημα σωστά, μπορούν και άσχημα Και το σύστημα δεν λειτουργεί όντως καλά. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε όμως, να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος για να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν πάμε πίσω μια γενιά ή όπως μας είπε ο κύριος Ραφαήλ στην αρχή, την αρχή της νομοθεσίας κατά του πλησίματος, το πλήσιμο γινόταν ε, ως κάτι δεδομένο διότι δεν έθεταν προβλήματα στους πελάτες τους και ερωτήσεις, δεν ρωτούσαν από πού είναι τα χρήματα και τι θα τα κάνουν. Η ρύθμιση κατέληξε τελικά να εξαφανίζει την αξία αυτής της διαδικασίας, έγινε θέμα χαρτιών. Αυτό δεν είναι καθε αυτό κακό ούτε και αυτό. Αλλά δεν μας λέει τι συμβαίνει. Και με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν υποτιμώ το ύψος των κεφαλαίων και συναλλαγών που διεκπεραιώνουν οι τράπεζες και για τη διαδικασία καταπολέμησης του πλησίματος. Αλλά αν και μόνο ένα τμήμα του κάθε χρόνο δινόταν στις διώξεις θα είχαμε πολύ αποτελεσματικότερες κυρώσεις. Δεν ζητάω νέα νομοθεσία. Ούτε καν νέες νομοθεσίες. Αλλά θέλω να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι αυτή η διαδικασία και ποιες είναι οι ευθύνες του καθενός μας για τη διευκόλυνσή τους ή για την παρεμπόδισή τους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και η κυρία προηγουμένως από τη Νομοσπονδία των Τραπεζών, οι τράπεζες είναι υπεύθυνες, το είπε με κάποια περηφάνεια, ευθύνονται για 80% αυτών των δοσοληψιών. Ναι, και κάνουν και αναφορές, ναι, αλλά δεν κάνουν τίποτα στις αναφορές αυτές, δεν τις κάνουν τίποτα. Οι τράπεζες ευθύνονται για 80% του προβλήματος επομένως. Αυτό σημαίνει. Και πρέπει οι αναφορές να μεταφράζονται σε βελτίωση των πραγμάτων. Αν μια τράπεζα, ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να βοηθήσει κυρία Πρόεδρε τη συζήτησή σας, την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο δικάστηκε ένας νεαρός Νιγηριανής καταγωγής που δούλευε σε μια τράπεζα τη UBS και που είχε χάσει 1,5 δισεκατομμύριο λίρες για την τράπεζα αυτή. Κόντεψε δε να τη ζημιώσει κατά 7,5 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι τεράστια ποσά. Αν ήταν τόσο απλό να ξεπληθεί τέτοιος όγκος χρημάτων, τότε κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα. Και ποιοι είναι καλύτερα σε θέση να το καταλάβουν και να αντιδράσουν. Το Ευρωπαϊκό. Με όλο το σεβασμό που οφείλω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πιστεύω ότι μεταξύ σας υπάρχουν άνθρωποι που είναι μαθηματικοί και traders και καταλαβαίνουν πώς δουλεύει η χρηματαγορά Κανένας εθνικός πολιτικός που, να τον, που έχω ποτέ γνωρίσει δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει εκεί μέσα. Να υποθέσει κανείς λοιπόν ότι εσείς μπορείτε να βρείτε την απάντηση είναι με όλο το σεβασμό που σας οφείλω λίγο φαντασιώδες. Αυτό που μπορείτε να αναμένετε είναι ο τομέας στον οποίο λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι να αριθμιστεί. Κυρία Πρόεδρε, αναφέρατε την περίπτωση του τράπεζας Μπάρκλεϊ που έδωσε σε έναν οικοσάρι ένα δάνειο ενός εκατομμυρίου ευρώ που βασικά χαρίστηκε, ήταν απάτη. Τέτοια γίνονται πολλά κάθε μέρα. Και ποιος ζημιώνεται, η Barclays και η μετοχή της. Αλλά μάλλον υπάρχει και ασφάλεια και αντασφάλεια. Γι' αυτό υπήρξε τέτοια ορμή για τα παράγωγα, για να δημιουργηθεί επικίνδυνο χρέος το οποίο να μπορεί να μεταπολιθεί και να αποβεί σε κέρδος. Όσο πιο επικίνδυνο τόσο πιο επικερδές. Εδώ υπάρχει ένα βιβλίο που γράφτηκε 3-4 χρόνια πριν που λέγεται Fool's Gold που δείχνει πώς ακριβώς δουλεύουν τα πράγματα. Αν οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να πάρουν τέτοιο βαθμό κινδύνου να αναλάβουν καθώς και τα έθνη και οι φορολογούμενοι, τότε πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς να ανατραπεί αυτό το φαινόμενο. Η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί καταρχήν στους μεσάζοντες. Οι χρηματοπιστωτικοί μεσάζοντες δεν είναι μόνο τράπεζες, κυρίως μεν τράπεζες, γιατί από αυτές περνάνε όλες οι ροές χρημάτων, αλλά ρητά λέω ότι φταίνε και δικηγόροι που δεν καταγγέλουν τις ύποπτες δοσοληψίες. Ξέρουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμιά πρόοδο και εγώ δικηγόρος είμαι και ευθύνομαι για τις δραστηριότητες των πελατών και πελατησών μου. Αν αυτοί και αυτές έχουν ύποπτες δοσο, κάνουν ύποπτες δοσοληψίες, έχω και εγώ ευθύνη. Και δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να το πούμε ρητά στους δικηγορικούς λόγους, ότι πρέπει να πείσουν τα μέλη τους ότι έχουν ευθύνη. Το ίδιο ισχύει και για, τις άλλες, για τα άλλα επαγγέλματα που μπερδεύονται με αυτές τις δοσοληψίες. Και αυτοί είναι οι μεσάζοντες. Όλοι αυτοί έχουν ευθύνη. Και πρέπει ο καθένας να αλλάξει νοοτροπία και να γνωρίζει πώς ο ίδιος κάνει κάτι για να διορθωθεί το πράγμα. Η τράπεζα που δεν εξετάζει καθώς πρέπει μία δοσοληψία επικίνδυνη, τι κάνει, τίποτα σχεδόν. Μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείε αναλαμβάνει η ευθύνη, γιατί εκεί υπάρχει νομοθεσία και είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς στα δικαστήρια ότι θα πει το ανώτατο δικαστήριο για αυτά τα πράγματα και τους υποστηρίζουν και οι δικηγόροι και οι δικαστές. Επιβάλλουν πολύ ψηλά πρόστιμα σε τράπεζες ευρωπαϊκές ή άλλες για τέτοιες εγκληματικές δοσοληψίες. Μερικές είναι πράγματι εγκληματικές, άλλες απλώς κατηγορούνται ως εγκληματικές αλλά αυτό αρκεί για να τις καταδικάσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εγώ ως Ευρωπαίος το θεωρώ πολύ αρνητικό στον κόσμο μόνον οι Ηνωμένε Πολιτείε να επιδίδουν ευθύνη στις τράπεζες για τέτοιες επικίνδυνες δοσοληψίες. Είναι πολύ σημαντικό και οι Ευρωπαίοι που παίζουν σημαντικό ρόλο ως ενδιάμεση χρηματοπιστωτέ να αποδώσουν και αυτοί ευθύνες Άλλο παράδειγμα. Η τράπεζα UBS που σας έλεγα επέτρεψε σε αυτόν τον trader της να τη ζημιώσει 1,5 δεκατομμύριο λίρες. Και το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ήταν γελίο. Είμαστε έτσι αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάρβερ. Ας μην ε, ξεχνάμε και το ρόλο των συμβολιογράφων ε, και των δικηγόρων αλλά και των συμβολιογράφων. Ε, μπορούμε νομίζω να μιλήσουμε για μια γκρίζα ζώνη που υποστηρίζει το οργανωμένο έγκλημα και διευνοεί τη διαφθορά και το ξέπλυμα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρλο Βαν Χιούκελο, ο οποίο είναι εκπρόσωπο τη Ευρωπόλ, ο οποίο θα μα μιλήσει για την επιχείρηση Αθηνά και για τι γενικέ μετακινήσει μετρητών, σε ένα στοιχείο για την πρόληψη τη νομοποίηση παράνομων εισόδων. Αν μπορείτε σύντομα, παρακαλώ να μα εξηγήσετε τι είναι η Europol και τι κάνει, για να μα ακούσουν και οι μαθητέ που είναι εδώ στην αίθουσα. Thank you, Mrs. Chairperson. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να σας παρουσιαστώ. Λέγομαι Κάρλο Βαν Χιούκελο και είμαι επικεφαλής ε, του ε, τμήματος ε, για το οικονομικό έγκλημα στη Γεροπόλ, η οποία είναι η υπηρεσία επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διευκολύνει και υποστηρίζει τα κράτη-μέλη ή τις διοκτικές αρχές στην καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος σε όλες τις μορφές. Θα δράξω την ευκαιρία να σας μιλήσω για δύο ζητήματα. Καταρχήν, το φαινόμενο ε, το ε, αποστολής χίδιν μετρητών που αυξάνεται συνεχώς και επίσης θα αναφερθώ στο ζήτημα ε, στο ε, χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Όπως σας ε, είπα, η κοινότητα διοκτικών αρχών είδε την τελευταία δεκαετία σημαντική αύξηση ιδίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λαθρέας ε, μετακίνησης ε, μεγάλων ποσών μετρητών που υλικά μεταφέρονται με κάθε είδους μεταφορικού μέσου, για σοδού οδού, με το τρένο, με το αεροπλάνο Υπάρχουν κάποιες εξωτερικές κινητήριες δυνάμεις που οδήγησαν ε, σε αυτή την ε, αύξηση του φαινομένου. Το 2002 είχαμε την εισαγωγή του ευρώ και του ευρώ και ε, κυρίως τα μεγάλα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ που διευκόλυναν την ηλική μεταφορά και την ανταλλαγή ε, παράνομων ποσών μετρητών. Ε, Παραδείγματο χάρη, να σα δώσω μια ιδέα, χρειάζεται σε ευρώ μόνο το ένα 8 του όγκου ε, σε σχέση με τα αμερικανικά δολάρια. Βλέπετε λοιπόν το πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί κανείς χαρτονομίσματα υψηλής αξίας σε ευρώ προσθέτω στο ευρώ γενικά ήταν ε, ένα νόμισμα σταθερό και γενικά αποδεκτό σε όλο τον κόσμο με σχετικά χαμηλή έκθεση στον πληθωρισμό. Ένα τρίτο, ένας τρίτος και πιο σημαντικός λόγος είναι ε, η Παγκόσμια Διάταξη κατά του ξεπλήματος βελούμικου χρήματος για να αποτρεπεί η κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για το σκοπό της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων έγινε κατά κάποιο τρόπο θύμα της επιτυχίας του. Δεν είναι η ηλίθιοι γενικά οι εγκληματίες και συνειδητοποίησαμε ότι για να μην τους βρουν ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούν όποτε μπορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα γιατί υπάρχει κάτι όπως αυτές οι εκθέσεις για τις ύποπτες συναλλαγές, οι STR, που επιτρέπουν ε, στις αρχές να ενημερώνονται όταν γίνονται κάποιες ύποπτες συναλλαγές μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης, ε, κάτι τελευταίο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, ως ένα βαθμό αυτό συνίστα μια ανομαλία κατά κάποιο τρόπο Μέχρι σήμερα υπάρχει απουσία κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να προβλέπει την υποχρέωση να υποβάλλονται αναφορές για εσωτερικά, εσωτερικές μετακινήσεις μετρητών ε, πάνω από 10.000 ευρώ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι πάνω από 10.000 ευρώ το ποσό που κουβαλάει κανείς ε, πρέπει να το αναφέρει σύμφωνα με τον κανονισμό 1889. Όμως σε περισσότερα, στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις μετρητών διασυνοριακά αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η τρίτη οδηγία κατά τη νομοποίηση παράνομων εσόδων υποχρέωσε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τα απαραίτητα νομικά μέτρα για να απαγορεύσουν τη χρήση των μετρητών για την ε, αγορά αγαθών. Ε, πρώτον αλλά όταν κάποιο ε, κουβαλά ε, μετρητά μέσα και τα φέρει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε κατά μέσο όρο 83.000 ευρώ αξία δηλώνεται κάθε φορά δεν υπάρχει μια τέτοια απαγόρευση και επομένως είναι κάπως δύσκολο να εξηγηθεί αυτό. Λόγω του φαινομένου αυτού που έχει καταστεί εμφανές τη τελευταία δεκαετία υπήρξε μια σειρά επιχειρήσεων που στήθηκαν ε, στο πλαίσιο της ομάδας συμβουλής του νόμου στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, προκειμένου να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Τρεις συνεχείς προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργάνωσαν την επιχείρηση Αθηνά, μια κοινή τελωνιακή και αστυνομική επιχείρηση προκειμένου να εντοπιστούν μετρητά και όπου ήταν δυνατό να κατασχεθούν. Η Προεδρία της Δανίας ε, νωρίς το 2012 ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει την ε, τρίτη τέτοια επιχείρηση, αλλά η Ευρωπόλ πρότεινε μια σχετικά διαφορετική προσέγγιση. Εμείς προτείναμε μία φάση, ένα στάδιο προεπιχειρησιακό που συνίστατο σε μία ανάλυση των κινδύνων και πρόκειψαν δύο πλεονεκτήματα από αυτό. Καταρχήν, μας επέτρεψε να στοχεύσουμε καλύτερα ε, τους ε, ε, μηχανισμούς που χρησιμοποιούσαν οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών κατά την ίδια την επιχείρηση και αυτό ε, δείχνει ότι ήμασταν αρκετά επιτυχείς ως προς την ε, σκοπιά αυτή Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ε, αυξήθηκε ο ρυθμός ε, των κατασχέσεων 600%. Ένα δεύτερο όφελος ε, που προέκυψε είναι επίσης εξίσου σημαντικό και είναι το εξή ότι για πρώτη φορά είχαμε συνολικές στρατηγικές πληροφορίες που μας επέτρεψαν να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο του προβλήματο, το πεδίο του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς του, που διέπουν το φαινόμενο αυτό. Τα κύρια πορίσματα του προεπιχειρησιακού σταδίου δεν θα σας τα αναφέρω εις βάθος, αναλυτικά, γιατί μπορείτε να διαβάσετε την παρουσίαση, θα τη διαθέσω στη συνέχεια. Όμως, τι μάθαμε. Ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι που μας επέτρεψαν να... πολλοί δρόμοι μας επέτρεψαν να επιτρέψουμε μας επέτρεψαν να, να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας εκεί, σε αυτές τις οδούς που χρησιμοποιούνταν ε, για την εμπορία μετρητών. και επίση ε, είδαμε και κάτι ξεθαύμαστο, όπως παραδείγματο χάρη, ότι ακόμη και το Μάρκο, ε, το γερμανικό, που δεν κυκλοφορεί πλέον ως νόμισμα, εξακολουθεί να κυκλοφορεί παρανόμως. Επίσης, βλέπετε εδώ κάποιες μεθόδους να κρύβουν τα μετρητά. Μοιάζουν πάρα πολύ με την εμπορία κοκαίνης και ναρκωτικών. Βλέπουμε εδώ κάποια παραδείγματα. Βλέπετε τι συναντήσαμε, πώς είχαν κρύψει τα μετρητά και πάει και πολύ μακριά. Μέχρι και κάποιοι να καταπίνουν μέχρι 35 προφυλακτικά που είχαν, τα είχαν γεμίσει με μετρητά. Βλέπετε λοιπόν πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι λαθρέμποροι. Κάποιος μάλιστα συνελήφθη να έχει στο στομάχι του 14 ράβδους χρυσού. Η κάθε μία από αυτές διηγήσε 100 γραμμάρια. Φανταστείτε να το καταπιεί κάποιο και να το βάλει αυτό στον οργανισμό του. Αλλά έχουμε αποδείξει ότι αυτό έχει συμβεί πάνω από μία φορέ. 26 χώρε μας έδωσαν στοιχεία προκειμένου να με δυσκολύνουν να κάνουμε μία ανάλυση βάση κινδύνων και στο πραγματικό ε, στάδιο ανάπτυξης τη επιχειρήση. 38 χώρε συμμετείχαν και πάλι δεν θα πω σε λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα και τα αριθμητικά στοιχεία. Αν σας ενδιαφέρει, ευχαρίστως ε, θα σας διαθέσω τα στοιχεία αυτά. Παρ' όλα αυτά, τι είναι σημαντικό. Να δούμε το συνολικό αποτέλεσμα σε σχέση με τα ποσά που μπαίνουν και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μετρητά και Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Μιλάμε εδώ ετησίως για μια συνολική αξία τουλάχιστον 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσά που επιτυχώς κατάσχονται είναι 155 εκατομμύρια ευρώ. Το ότι κατάσχονται αυτά τα χρήματα σημαίνει ότι αυτός που τα κουβαλούσε δεν κατάφερε, μάλλον απέτυχε να τα δηλώσει σύμφωνα με την υποχρέωση που θεσπίζει ο κανονισμός 1889 του 2005. Φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο το ποσό αυτό και μπορώ να σας πω ότι κατόπιν ανάλυσης έχουμε τρεις φορές περισσότερα μετρητά που εγκαταλείπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από όσα μπαίνουν. Οι διαδοχικές επιχειρήσεις μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε κάποια συγκεκριμένα pattern, κάποια συγκεκριμένα μοντέλα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι ένα ποσό 430 εκατομμυρίων δολαρίων και 10 εκατομμυρίων ευρώ ουσιαστικά μεταφέρθηκε, διαμετακομίστηκε από την Ουκρανία μέσω επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. χρησιμοποιούν την αποκαλούμενη συλλογική δήλωση. Δηλαδή έρχονται με ένα λεωφορείο, περνάνε τα σύνορα και ο οδηγός δηλώνει συλλογικά τα μετρητά που κουβαλούν οι επιβάτες του λεωφορείου. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια πραγματική και χρήσιμη χρήση της ε, υποχρέωσης του κανονισμού 1889. Τα μέτρα που λάβαμε. Ως προς την εκμετάλλευση αυτών των πληροφοριών. Δυστυχώς ε, δεν ε, ήταν κατελοκληρωμένο καθώς οι εξωτερικοί μας εταίροι δεν ήθελα να συμβάλλουν στις προσπάθειες, καθώς ε, είπαν ότι αυτές ε, οι ταμιακές ροές ε, σχετίζονταν με κάποιους εμπόρους και θεωρούσαν ότι δεν ήταν σοβαρό αδίκημα. Με κάποιους εμπόρους βαποράκια σχετίζονταν λοιπόν και δεν θεώρησαν όταν σοβαρό δίκημα. Ε, λοιπόν, με, για τη μεταφορά ε, κάποιων ε, ποσών από τα σύνορα χρησιμοποιούνται κάποιοι δείκτες κόκκινη σημαία ε, της ε, Task Force και υπάρχουν ε, κάποιες δυσκολίες να ε, τεθούν σε εφαρμογή οι δείκτες αυτές, όταν ε, κατατύχει τελικά ε, αυτοί οι courier, αυτοί που μεταφέρουν τα μετρητά, τα δηλώνουν, δεν έχουν εξουσία να κατάσχουν και να δημεύσουν αυτά τα χρήματα. Κάποιος δηλώσει στο αεροδρόμιο ένα μεγάλο ποσό, αλλά πετάμε μια διασυνοριακή πτήση. Πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει τη φύση της συναλλαγής. Επίσης έχουμε τεράστιες δυσκολίες ε, να επαληθεύσουμε και να αποδείξουμε κάποιες ε, ψεύτικες, ψευδείς ή ε, μη πλήρης ή ανακριβείς πληροφορίες. Επίσης, να βρούμε τις ενδείξεις ότι αυτά τα ποσά σχετίζονται με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα το χαρτονομίσμα των 500 ευρώ. Θα γνωρίζετε κάποιοι και είναι γενικώ γνωστό το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΣΟΚΑ, η Υπηρεσία καταπολέμηση του Σοβαρού και Οργανωμένου Κλίματος, βάσει του ότι έχουν στρατηγικές πληροφορίες ε, ότι κατά 95% το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ χρησιμοποιούνταν κυρίως από το οργανωμένο έγκλημα, έλαβαν κάποια διοικητικά μέτρα, η υπηρεσία αυτή έλαβε κάποια διοικητικά μέτρα για να απαγορεύσει ε, την κυκλοφορία αυτού του χαρτονομίσματος στην επικρατειά του. Δεν θα πήγαινα τόσο μακριά όσο να πω ότι τα μεγάλα χαρτονομίσματα απλώς διευκολύνουν το οργανωμένο έγκλημα, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εγχείρημα να εξετάσουμε αν αιτιολογείται οικονομικά η ύπαρξη τέτοιων χαρτονομισμάτων. Υποθέτω ότι πολλοί από εσά, όπως και εγώ, σχεδόν ποτέ δεν ε, συναντούν ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Παρόλα αυτά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων χαρτονομισμάτων σε κυκλοφορία. Προκειμένου λοιπόν να αξιολογήσουμε κατάλληλα την κατάσταση, μας ζητήσαμε μία αναλογία που να, μας που να μας επιτρέπει να κάνουμε μία συγκριτική μελέτη μεταξύ των τριών μεγάλων νομισμάτων που γνωρίζουμε σε αυτό το τμήμα του κόσμου, δηλαδή το αμερικανικό δολάριο, την λίρα και το ευρώ. Και δεν έχει κανένα νόημα απλώς να συγκρίνουμε τα ποσά που είναι στην κυκλοφορία, Απλώς λοιπόν ε, αναπτύξαμε μία αναλογία που αιτιολογείται επιστημονικά, που είναι ο όγκος ενός συγκεκριμένου νομίσματος σε κυκλοφορία, σε χαρτονομίσματα, σε τραπεζογραμμάτια, σε σχέση με το ΑΕΠ. Και το εγχείρημα αυτό μας έδωσε κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Γιατί όπως βλέπετε εδώ, ο όγκος των τραπεζογραμματείων στην Ευρωζώνη είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον όγκο των τραπεζογραμματείων σε αμερικανικά δολάρια που κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο. 7,59% του συνδυασμένου ΑΕΠ της Ευρωζώνης είναι σε κυκλοφορία σε τραπεζογραμμάτια από τα οποία 2,53% σε χαρτονομίσματα 500 ευρώ είναι σε κυκλοφορία και σε σύγκριση με τα αμερικανικά δολάρια υπάρχει σημαντική διαφορά. Και επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ε, το υψηλότερο χαρτονόμισμα σε αμερικανικό δολάριο είναι το χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων, ενώ σε ευρώ έχετε και ε, χαρτονόμισμα των 100, των 200 και των 500 ευρώ. Και ξέρετε ότι και τα τρία κοστίζουν, αξίζουν πιο πολύ από ένα χαρτονόμισμα 100 δολαρίων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει εδώ κάτι και σύντομα θα καταλάβετε ποιο είναι το ζήτημα σε σχέση με το χρητονομίσμα των 500 ευρώ. Όταν σας ανέφερα ότι το εισόδημα το 2008 στο κράτη-μέλη ήταν 226 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, πρέπει να κατανοήσετε ότι η έκδοση των χρημάτων και το εισόδημα που γεννά είναι επίσης ένα σημαντικός ε, παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αξιολογείται η χρησιμότητα ε, του να κυκλοφορούν νομίσμα, χαρτονομίσματα με τόσο υψηλής αξία. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε τρεις παρεμβάσεις ε, στο ύψος ε, ε, των προσδοκιών της Επιτροπής μας. Να κάνω κάποιες γρήγορες ερωτήσεις. Το θέμα που συζητήσαμε αφορούσε τις περιφέρειες που δεν συνεργάζονται για την καταπολέμηση του φαινομένου της νομοποίησης σε οδών. Αναφέρθηκαν και η Κύπρος, η Σιγκαπούρη, το City του Λονδίνου, έχουν κεντρικό ρόλο σε σχέση με αυτό το φαινόμενο. Να σας ρωτήσω και τους τρεις. Είναι δυνατό να αξιολογήσουμε, να μετρήσουμε με συγκεκριμένους όρους πώς το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με τα όσα συμβαίνουν σε αυτές τις περιοχές. Ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος ε, της κατάσχεσης. Όμως, παραδείγματος χάρη, είχαμε και το κελιό του Ντουίσμπουργκ. Εκεί χρησιμοποιήθηκε στη Γερμανία για να υπάρξει ε, ουσιαστικά μια ανανέωση του συστήματος και για την Ελβετία αναφέρθηκε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τρομοκρατίας και ξεπλήματος και επίσης μιλήσατε και για το επίπεδο κινδύνου των τραπεζών. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει κοινή γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναχέτηση αυτού του φαινομένου και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και μια συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να αξιολογήσουμε τους τραπεζικούς κινδύνους και να επιτεθούμε από κοινού στο φαινόμενο αυτό. Και τέλος κάτι να πω σε σχέση με την ε, παρέμβαση του Βαν ε, Ελκελόμ, του εκπροσώπου της ε, Europol οι πόροι επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα project, αξιολογήσιμα που τέθηκαν σε εφαρμογή ε, με συνεργασία τελωνιακών και αστυνομικών αρχών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σήμερα είναι και σημαντική ημέρα γιατί καταγράψαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι το πρωταρχικό ζήτημα είναι να προβλέψουμε μέτρα, εργαλεία αποφασιστικά όπως είναι η δέσμευση. Γιατί με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και σε σχέση με την συνταστηριότητα των νομιμοποίησης παράνομων εισόδων. Μάλιστα, ευχαριστώ κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους τρεις για τις παρεμβάσεις τους που ήταν τόσο ενδιαφέρουσες. Κύριε Φίντλερ. Μιλήσατε για κατασχέσεις και για την απογοήτευση που έχετε στον αγώνα σας λόγω της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών με διαφορετική νομοθεσία ή με την νομοθεσία που ισχύει σε σύνδεση, σε σύγκριση με το σχέδιο οδηγίας της Κομισιόν. Το πρωί μιλούσαμε με τον εκπρόσωπό της και το θίξαμε και αυτό σε μια άλλη επιτροπή, όχι στη δική μας. Το συζητάμε δε συνεχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι είναι πολιτικό το πρόβλημα όπως είπατε, αλλά δυστυχώς η κυβέρνησή σας και η δική μου, το κράτος σας και το δικό μας, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, είναι χώρες που δεν περνούν στην επόμενη φάση. Δεν υπάρχει θέληση. Η Γερμανία, η Γαλλία, λυπούμε γι' αυτό, μας θέτουν ιδιαίτερα νομικά προβλήματα. Οι δικοί μου μου λένε όχι, είναι πολύ πολύπλοκα όλα αυτά, δεν θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω και να επιτρέψουμε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αν δεν έχει υπάρξει καταδίκη ή αν έχει κανείς πεθάνει ή αν είναι άρρωστος, τότε δεν μπορεί να γίνει η κατάσχεση. Ή ακόμη κι αν δικάζεται και ανάλογο πρόβλημα από ό,τι ξέρω υπάρχει και με Στη Γαλλία απαντώ μα αλλάξτε αυτή την νομοθεσία, αλλάζουν οι νόμοι. Και στη Γερμανία μπορούν να αλλάξουν, παντού μπορούν να αλλάξουν. Αλλά δεν υπάρχει πολιτική θέληση και αν δεν υπάρχει πού θα πάμε. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη θέληση στεναρή στο Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό υπάρχει, αλλά όχι τόσο πολύ στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι που λείπει. Καλό είναι λοιπόν που το είπατε και εμείς οι βουλευτέ πρέπει να πιέσουμε για να γίνει κάτι. Κύριε Βανόκελομ, μου άρεσε πολύ η παρέμβασή σας, πράγματι τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ αναρωτιέται κανείς γιατί υπάρχουν μόνο για να διευκολύνουν τη μαφία που έχει να περάσει πολλά χρήματα. Τα 500 ευρώ νομίζω χρησιμεύουν για να μεταφερθούν τεράστια ποσά βέβαια, όχι για τους ε, ψιλικατζίδες. Αλλά Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσεως εγώ κατοικώ στην περιοχή των Βοσγίων κοντά στο Στρασβούργο σε ένα νομό που υποφέρει πολύ και 50 ευρώ ακόμη χαρτονόμισμα δύσκολα χαλιά, χαλάει σε μερικά μαγαζιά όπως στο Αρτοποιείο, στο μπακάλικο, στο μανάβικο. Φανταστείτε με 500 τι γίνεται. Δεν μπορώ να φανταστώ σε τι κύκλωμα κυκλοφορούν αυτά τα χαρτονομίσματα. Μόνο μαφιόζικο δίκιο έχετε. Υπάρχει ιδέα να αλλάξουν οι κοπή των χαρτονομισμάτων στην Ένωση. Ελπίζω να καταργηθεί το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ γιατί απλώς διευκολύνει την μαφία. Ευχαριστώ. Α, πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νιούτον Ντάμπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ε, τρεις ε, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Προς τον κύριο Φίτλερ είπατε κάτι πολύ ε, σωστό. Το έγκλημα στοιχίζει περισσότερο από την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλης στα κράτη-μέλη να γίνουν τα απαραίτητα. Εμείς ελπίζουμε ότι η δική μας έκθεση όταν θα δημοσιευτεί το καλοκαίρι ε, θα περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία που θα δείχνουν το πρόβλημα και έτσι λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη θα πιεστούν να λάβουν μέτρα. Μήπως λοιπόν έχετε στοιχεία να μας πείτε ποιο ακριβώς είναι το κόστος πίσω από αυτή τη θαυμάσια δήλωση που κάνατε. Ε, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποια στατιστικά δεδομένα. Ε, τώρα προς τον κύριο Κάρβερ ε, και πάλι ψάχνω να βρω στοιχεία. Εσείς είπατε οι παράνομες ροές αυξάνονται εκθετικά. Έχετε και εσείς στοιχεία. Και αυτό θα ήταν χρήσιμο. Επίσης είπατε πολύ σωστά ότι οι ευρωβουλευτές δεν είναι ειδικοί στις αγορές χρήματος. Εμείς ε, γενικά ασχολούμαστε με όλα, όπως και οι εκπρόσωποι του Κογκρέσου. Απλά προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Μήπως λοιπόν να ε, μας ε, παραπέμψετε σε ειδικού για την αγορά χρήματος που ίσως να τα ξέρουν καλύτερα και να μας πούνε μια φόρμουλα, έναν τύπο που να πρέπει να συμπεριλάβουμε και προς τον κύριο Βαν Χόκελεν. Ζητώ συγγνώμη που δεν ξέρω, αλλά μπορείτε να μου επενθυμίσετε γιατί χρειαζόμαστε ένα νόμο για να εμποδίσουμε τους ανθρώπους ε, να μεταφέρουν μετρητά. Γιατί να υπάρχει τέτοιου είδους νόμος απλά και μόνο για να αντιμετωπιστούν οι εγκληματίες, αυτός είναι ο λόγος. Και ε, όπως είπε και η Βερονίκ, θα πρέπει να προτείνουμε να καταργηθούν τα πεντακοσάρικα. Ε, αυτό θα σας βοηθούσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μποργκέζε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με, την, με το γερμανό αστυνομικό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Μετά την σφαγή στο Ντουίσμπεργκ, η αστυνομία στη Γερμανία κατόρθωσε μήπως ε, να ε, εντοπίσει την οικονομική διείσδυση της Ιταλικής ε, μαφίας στη Γερμανία. Το κατόρθωσε αυτό η αστυνομία. Και μία άλλη ερώτηση. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού. Ποιοι είναι οι τομείς όπου ε, αναπτύσσονται κυρίως δραστηριότητες όχι μόνο διείσδυση αλλά και επενδύσεων ε, και ε, δραστηριότητε ξεπλήματος. Όσον αφορά τον εκπρόσωπο της ε, Transparency International, θέλω να τον επενέσω για το ότι υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του City του Λονδίνου σε αυτό το διεθνές και παγκόσμιο πλαίσιο των ε, γκρίζων δραστηριοτήτων ε, του, της παγκόσμιας κοινωνίας ε, του χρήματος. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τη σχέση ανάμεσα στη διείσδυση κεφαλαίων, εγκληματικών κεφαλαίων και στις χρηματικές κερδοσκοπίες, η κρίση δηλαδή, όλα αυτά που προκάλεσαν την παγκόσμια κρίση. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο. Και αν ναι, κατά τις αναλύσεις, τι ακριβώς έχει προκύψει. Και όσον αφορά στον προστατευτικό ρόλο της ε, City απέναντι σε αυτά τα ε, ανέγγιχτα κυκλώματα, ποια είναι τα αποτελέσματα των ε, προσπαθειών να ε, μπορέσει κανείς να μπει σε αυτό το χώρο. Όσον αφορά τη Europol, αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ήταν αυτό που είπατε, που δώσατε ιδιαίτερη σημασία στην κυκλοφορία των πεντακοσάρικων. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε καλύτερα για τις χώρες όπου έχετε εντοπίσει κυρίως μεγάλες ποσότητες τέτοιων χαρτονομισμάτων. Και τι είδου ε, δραστηριότητες ε, ανάλυσης, ποιες αναλύσεις κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει αρκετά στοιχεία που να αφορούν σε αυτό το φαινόμενο. Τι ρόλο παίζει. Και τέλος, ε, όσον αφορά τις αναλύσεις σας για την φαιά ζώνη της διείσδυσης και των ε, δραστηριοτήτων και ξεπλήματος ε, των εγκληματικών οργανώσεων, Πολύ σωστά μιλήσατε για τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το τραπεζικό σύστημα και οι επαγγελματίες. Όμως Μόνο αυτά είναι τα κανάλια που υπάρχουν, αποκλειστικά αυτά και μόνο. Ή μήπως, να το πω αλλιώς, η ευθύνη ε, αφορά μόνο όσους ε, διευθύνουν τις ε, τράπεζες και αυτούς τους οργανισμούς, η ευθύνη βαρύνει αυτούς μόνο ή μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ε, αυτή η προστασία οτι αυτη η εκείνη που εμποδίζει να ε, ρηχθεί φως ε, σε αυτές τις ε, δραστηριότητες. Ας πούμε, Bilderberg ή διεθνής, μασον, διεθνής μασονία αυτοί έχουν ε, ειδικό ρόλο στο να προσφέρουν προστασία μέσα από τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις. Δις μέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσο πιο σύντομα μπορώ θα κάνω κάποια σχόλια. Τα δύο να πάνελ ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Και Ας ξεκινήσουμε από το θεμελιώδες, γιατί το θεμελιώδες ε, είναι να περιγράφουμε τα φαινόμενα. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνουμε στο ουσιαστικό και αυτό είναι το πώς θα απαντήσουμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Η συζήτηση είναι ενδυμική, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η καταπολέμηση του εγκλήματος ε, πάντοτε σύσταται σε δύο θέματα στην καταπολέμηση κατά της ε, παράνομης ε, χρηματοδότησης και κατά της νομιμοποίησης παράνομων εισόδων και κατά του εγκλήματος αφενός και αφετέρου η προστασία των προσωπικών δεδομένων για των προσωπικών ελευθεριών. Υπάρχουν ε, κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ε, δεχτεί επίθεση από τον τρόμο, αλλά και χώρες που βρίσκονται στην ε, αντίθετη κατάσταση και απαντούν σε αυτές τις προκλήσεις. Αυτό το σχόλιο το συνδέω με κάτι που είπε ο κύριος Κάρβερ με τη μορφή μιας ιστορίας. Είπε και έχει δίκιο ότι δεν είμαστε ειδικοί στα παράγωγα, αλλά δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να είμαστε εμπειρογνώμονε στα χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Εμείς είμαστε νομοθέτε και ω νομοθέτε προσφεύγουμε σε εμπειρογνώμονε. Και αυτό που κάνουμε και το κάνουμε καλά σε αυτό τον οίκο είναι να εγκρίνουμε ή να απορρίπτουμε να εγκρίνουμε ή να απορρίπτουμε διεθνείς συμβάσεις σχετικές με χρηματοοικονομικές συναλλαγές διεθνείς. Εσείς πολύ καλά υπενθυμίσατε, γιατί εδώ, στο Βέλγιο, ξέσπασε το σκάνδαλο της SWIFT, δηλαδή της μαζικής αποστολής δεδομένων, σχετικά με διεθνείς ε, τραπεζικές συναλλαγές. Και αυτό οδήγησε σε μια δύσκολη κατάσταση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό ε, είχε να κάνει με μια σύμβαση αμφίσιμη που τελικά εγκρίθηκε και από το Κοινοβούλιο και έδωσε μια αρμοδιότητα στη Europol που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ως κοινή αρχή ελέγχου τη στιγμή που ελέγχει και φιλτράρει όλη αυτή την διαβίβαση των δεδομένων. Και να ολοκληρώνω στι Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι μια χώρα η οποία δέχεται επίθεση από τον τρόμο και από το ξεπλημένο έχουν ένα σύστημα που λέγεται TFTP. Έχουν ένα πρόγραμμα για να προστατευτούν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πλήθος νομοθεσιών στα κράτη-μέλη, κανονισμούς, οδηγίες. Έχουμε εντοπίσει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όμως δεν έχουμε μία ισχυρή TFTP. Και, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η απάντηση, η ουσιαστική και που έρχεται μετά από το θεμελιώδες. Αυτό που έρχεται αφού εντοπίσουμε το πρόβλημα. Αυτό που έρχεται αφού συζητήσουμε τα προβλήματα. Όταν, ε, ολοκληρώνεται, όταν ολοκληρωθεί η προσωρινή εργασία, του προσωρινό έργο αυτής της Επιτροπής, θα πρέπει κάτι να συνεισφέρουμε. Και σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα το απόγευμα, εγώ λέω το εξή. Ξέρουμε ότι ήδη έχει ασχοληθεί άλλη επιτροπή με αυτό το θέμα, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, κοινό πρόγραμμα προστασίας. Όχι μια κοινή φωνή, όπως λέγεται συχνά εδώ, αλλά ένα κοινό πρόγραμμα, δηλαδή ένα νομοθετικό μέσο κοινό. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δίας Δεμέρα. Και πάλι να δώσουμε το λόγο στους συζητητές μας. Έχετε πολύ πιο λίγο χρόνο, μόνο τρία λεπτά ο καθένας για να απαντήσετε. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Φίγκλερ. Das wird Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή, όλα σε τρία λεπτά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Η πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν να αποσωστικοποιήσουμε το πρόβλημα. Πόσο κοστίζει η συνεργασία μας με τα διάφορα κράτη. Δεν έχω μελέτες για αυτό το θέμα, δεν έχω. Αυτός που τις είχε δεν έφυγε αλλά από ό,τι ξέρω υπάρχει μια μελέτη αν δεν απατώμε, αλλά δεν μου έρχεται τώρα. Δεύτερο ερώτημα για την απογοήτευση που είχα εκφράσει προηγουμένως στην ομιλία μου. Είχα μιλήσει για την πολιτική εφαρμογή όλων αυτών. Ένα παράδειγμα που μπορεί να σας τα εξηγήσει όλα, πώς μπορεί μια πολιτική συζήτηση να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Έχουμε το εξή ε, πρόβλημα. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή είμαστε ομοσπονδιακό κράτο και μέσα στη Γερμανία. Και παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που ανησυχούν την κοινωνία γιατί εμφανίζονται πολύ περισσότερο από τα θέματα που συζητήσαμε εδώ. Και καταρχήν όπως σας είπα υπάρχει η ε, φαιά ζώνη. Στη Γερμανία, στα 16 κρατήδια, ε, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες πως οι αστυνομικοί παραδείγματος χάρη θα πρέπει να ελέγχουν ε, τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις διαδηλώσεις. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τι είδου προσόντα θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να είναι σαφές, να έχουν συμφωνήσει όλα τα πολιτικά κόμματα ότι πρέπει να ε, συμφωνούν για την ποσότητα, όπως σας είπα, τον αριθμό και τα προσόντα. Στην ε, αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ε, δεν υπάρχει αυτή η συνένεση και στα διάφορα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι λιγάκι περίεργο, αλλά με οδηγεί σε κάτι ε, το ότι ισχύει πάντα αυτό στη διαχείριση, δηλαδή υπάρχουν δύο αίτια. Είτε η αγάπη για το νέο είναι πολύ μεγάλη ή υποφέρει κανείς τόσο πολύ που να θέλει αλλαγή στο πολιτικό σύστημα. Στα κράτη-μέλη λοιπόν το βλέπουμε αυτό. Στην Ιταλία παραδείγματο χάρη, αν δούμε τις ρυθμίσεις που υπάρχουν εκεί, αυτές οι ρυθμίσεις υπάρχουν από την υπερβολική πίεση. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι όταν είναι συνδυτά τα προβλήματα, όταν τα συνειδητοποιούν οι πολίτες, βεβαίως είναι και σε θέση να επιφέρουν αλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, βλέπουμε ότι πολλοί δεν αντιμετωπίζουν την ε, πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν γίνεται συνδυτή για πολλούς. Τώρα, όσον αφορά αριθμούς και γεγονότα, ε, βεβαίως και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και αριθμοί που γνωρίζουμε, αλλά αυτό που μας λείπει κυρίως είναι η έρευνα. Εκείνο που γνωρίζουμε βέβαια είναι το εξής και αυτό το έχει πει η δική μας υπηρεσία. Το maximum που πιάνουμε είναι το 1%. Ούτε καν τους μισούς δεν πιάνουμε. Στη Γερμανία έχουμε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ που τα εξασφαλίζουμε κάθε χρόνο. Ε, αυτά όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι στη Γερμανία το ποσό που διακινείται είναι 15 δις. Και βλέπετε λοιπόν τα στοιχεία είναι πάρα πολύ συντηρητικά. 10 με 20 δις είναι το παράνομο χρήμα ε, στα διακινούμενα κεφάλαια. Ε, άρα δηλαδή οι αριθμοί είναι εντυπωσιακή. Το θέμα είναι, όπως σας είπα, ε, το τι κατορθώνουμε να πιάσουμε. Και εκεί δυστυχώς ε, ε, δεν, είμαστε, δεν, δεν σημειώνουμε επιτυχία. Στο Ντουισμπουργκ που θίξατε εσείς, η ερώτηση ήταν αρκετά ευρεία. Βεβαίως και γνωρίζουμε ότι η μαφία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον τομέα των ακινήτων, των σκουπιδιών. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι το θέμα των τυχερών ε, παιχνιδιών. Ε, αυτά είχα να σας πω. Ε, δεν είχα και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι κύριε Γιακολίνο. Ίσως δεν με καταλάβατε καλά. Δεν είπα ότι το σίτι του Λονδίνου είναι από τις μη συνεργαζόμενες περιφέρειες. Είπα ότι μάλλον είναι το μεγαλύτερο πλυντήριο χρημάτων στον κόσμο, πράγμα το οποίο οφείλεται απλώς και μόνο στο γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό μέρος του κόσμου. Υπάρχει δηλαδή εκεί μεγάλη ροή χρήματος και ένα τμήμα του πάντα είναι παράνομο. Χρόνια λέω ότι το City του Λονδίνου έχει ιδιαίτερη ευθύνη. Ως η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική, το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό μέρος του κόσμου και θα μπορέσει αν κάνει κάτι για να καταπολεμήσει το ξέπλυμα να ωφελήσει όλο τον κόσμο. Χαίρομαι γιατί η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το καταλαβαίνει αυτό και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι το θέμα θα το θίξει ως τμήμα του προγράμματός της όταν θα προεδρεύσει στο Z8 του χρόνου. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θέλει να επιδείξει ρεαλισμό και έλλειψη υποκρισίας και αλαζονίας ότι όλα είναι εντάξει στο Ηνωμένο Βασιλείο, γιατί δεν είναι. Δεν είναι χειρότερα τα πράγματα σε εμά από ό,τι αλλού, αλλά υπάρχουν αδυναμίες και οι αδυναμίες αυτές πρέπει να ταυτιστούν και να λυθούν. Δεν θα τις λύσουν οι κυβερνήσεις, ούτε το Αγγλικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να λυθούν από τους ίδιους εκείνους που διαπράττουν τις δοσοληψίες αυτές. Από τους μεσάζοντες δηλαδή. Αυτοί ξέρουν το σύστημα και αυτοί πρέπει να ενθαρρυνθούν και να πάρουν κίνητρα θετικά ή αρνητικά για να διασφαλίσουν ότι το σύστημα θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Αυτό ψάχνω εγώ. Αυτό ζητάω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνει σε κάθε χρηματοπιστωτικό κέντρο στην Ευρώπη. Με τον ίδιο βαθμό αναγνώρισης της πραγματικότητας χωρίς αλαζονία και με την επικοδομητική επιθυμία να αλλάξουν τα πράγματα. Αν δω τα κοινοβούλια βλέπω ότι παίζουν κυρίως πολιτικό και όχι απλώς νομοθετικό ρόλο. Υπάρχει πάρα πολύ νομοθεσία στον κόσμο και το μεγαλύτερο της μέρος δεν ωφελεί. Το πολιτικό όμως μήνυμα πρέπει να είναι ισχυρό δηλαδή να βασίζεται στην αναγνώριση των αδυναμιών για τις οποίες είμαστε και εμείς υπεύθυνοι και στην κατανόηση του πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικότερα. Όλοι οι ομιλητές το απόγευμα μίλησαν για το ότι χρειάζεται περισσότερο πιο αποτελεσματική συνεργασία. Αυτό ισχύει και εθνικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα τρομερά αναποτελεσματικό σύστημα αστυνομικών δυνάμεων που δεν πολύ συνεργάζονται. Άλλος συνάδελφος μίλησε για 200 τέτοια σώματα. Δεν γίνεται τίποτα έτσι. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία και συνεννόηση. Υπάρχει τρόπος. Θα ήθελα να πιστεύω ότι μερικά από τα μαθήματα που παίρνει το Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε ότι οι χρηματοπιστωτικές η αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει αποτύχει να ρυθμίσει τη λειτουργία του ΣΥΤΙ. Τώρα θα αλλάξει ο διευθυντής της, θα βάλουν τον ε, πρώην κυβερνήτη της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά ως πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας. Πρέπει να πειραματιστούμε και να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζονται καινούργια πράγματα αν καταλάβουμε το σύστημά μας ο καθένας, τότε μπορούμε και διεθνώς να συνεισφέρουμε περισσότερα. Σε ευρωπαϊκά βήματα ή σε ευρύτερα βήματα. Γίνεται αυτό, υπάρχουν τέτοια, τέτοιοι τρόποι, αλλά πρέπει να έρθουμε στο τραπέζι των συνεννοήσεων με πραγματική επιθυμία να πειραματιστούμε μαζί και επικοδομητικά. Ο κύριος σε αλλά πρέπει να ξέρετε ότι σε πέντε λεπτά αρχίζει εδώ συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Ορίστε. Θα περιοριστώ στο κατά πόσον θα ήταν καλό να that, but would be... να καταργήσουμε ορισμένες προτάσεις. Καλύτερο μου φαίνεται θα ήταν να ξέρουμε ότι κάθε χρόνο από την Νότια Αμερική έρχονται 2-3 δισεκατομμύρια ευρώ σε χαρτονομίσματα 200 ευρώ. Τι συμβαίνει εκεί. Τόσο πολλοί Ευρωπαίοι τουρίστες, 500 μάλλον ευρώ, τόσο πολλοί Ευρωπαίοι τουρίστες πάνε στη Λατινική Αμερική με τέτοια χαρτονομίσματα τόσο μεγάλα. Δεν καταλαβαίνω τι κρύβεται εδώ. Επίσης, υπάρχει και η βασική οικονομική αρχή ότι πρέπει τα χαρτονομίσματα να τα θεωρήσουμε ως οποιοδήποτε εμπόρευμα. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Αν έχουμε μεγάλη ζήτηση τότε μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας, δηλαδή τα έσοδα που έχουμε από την έκδοση χρήματος. Αν αναρωτηθείτε από πού προέρχεται η ζήτηση αυτών των μεγάλων χαρτονομισμάτων, τότε θα καταλάβετε, θα έχετε πολλές απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Τέλος, ποια χώρα εκδίδει το μεγαλύτερο αριθμό πεντακοσάρικων από τους αριθμούς που έχουμε από την ΕΚΤ που είναι από το 2007 φαίνεται ότι το 55% εκδίδονται από τη Γερμανία. Τέλος, αν θέλετε να καταργηθεί το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, θα ακούσετε αντιδράσεις που δεν φανταζόσασταν. Η κυρία Ματιέ ζήτησε το λόγο. Ένα ερωτηματάκι προς την Ευρωπόλ. Στη Γαλλία υπάρχει ανώτατο όριο και φαντάζομαι και στις άλλες χώρες που δεν μπορεί να ξεπεραστεί για τις πληρωμές σε χρήμα. Στο Βέλγιο τι ισχύει. Δεκαπέντε ευρώ. σε Λοιπόν, επειδή σίγουρα ε, είχατε λιγότερο χρόνο για να απαντήσετε από τις ερωτήσεις που σας ετέθησαν, αν θέλετε ε, μπορείτε να μας στείλετε με email τις ε, παρατηρήσεις. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά ήσασταν ε, και ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και απόλυτα ε, ξεκάθαροι, γιατί πολλές φορές ε, πολλοί υποβάλλουν ερωτήσει, αλλά οι απαντήση δεν είναι σαφής. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την διαθεσιμότητα που δείξατε. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους άλλους ε, ταχύτατα ε, ώρα Επόμενη συνεδρία στις 3 Δεκεμβρίου.